Okay, hello everyone. Καλό σας απόγευμα. Θα αρχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό Υγείας, ε, την κυρία Σωρίνα Πίντε, η οποία θα εκπροσωπήσει τον τομέα της υγείας στα πλαίσια της Προεδρίας και φυσικά εθιμοτυπικά μας επισκέπτεται για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες και τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ελπίζουμε να τα καταφέρετε μέχρι το τέλος της ε, θητείας. Για μας αυτό το θέμα είναι ύψης της σημασίας, η υγεία γενικότερα. Γι' αυτό και η επίσκεψή σας ήταν αναμενόμενη. Χωρίς να παρατείνω την εισαγωγή, θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρουμανική Προεδρία στον τομέα της υγείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να προωθήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα σε σχέση με τα ευεργετήματα υπέρ των ασθενών. Κατά την εντολή μας αυτή, κατά την Προεδρία, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρόσβαση στην υγεία για όλους τις πολίτες. Το πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας αφορά την ε, μικροβιακή αντίσταση, τον εμβολιασμό, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, την ε, κινητικότητα καθώς και την ψηφιακή υγεία. Όλα αυτά τα θέματα που προτείνει η Προεδρία είναι επίκαιρα ζητήματα για την βελτίωση των παροχών και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας αλλά και στον τομέα της πρόληψης. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ορισμένα βασικά στοιχεία του προγράμματος της Προεδρίας καθώς και τις δράσεις που θα θέλαμε να προωθήσουμε μέσα στα πλαίσια των στόχων μας. Σε σχέση με την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας, αυτό είναι το μόνο θέμα που απασχόλησε πρόσφατα την ΕΠΣΚΟ. Και η Ρουμανική Προεδρία θα προτείνει έναν κανονισμό για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας. Αυτή είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι τόσο οι ασθενείς όσο και τα συστήματα υγείας μπορούν να έχουν μία παγιωμένη ε, συνεργασία στον τομέα της υγείας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη πόλωση σε σχέση με τις συνέπειες αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας, όλες οι αντιπροσωπείες έκναν σκόπιμη τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό καθήκον, ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξει αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να επιτελεστεί πρόοδος. Η Ρουμανία θα σας μιλήσει για τις πρόοδους ε, με βάση το Συμβούλιο Θεμάτων Υγείας της 14 ε, Ιουνίου. Έχουμε προβλέψει πολλές συνεργασίες και η πρώτη έγινε στις 8 Ιανουαρίου ως προεδρεύουσα θα προσπαθήσω να είμαι ένας αμερόληπτος μεσολαβητής για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και διμερός με τους ομολόγους μου. Μία άλλη προτεραιότητα της Ρουμανικής Προεδρίας είναι η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Το θέμα της επωνομαζόμενης μικροβιακής αντοχής ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιφέρειες όπου υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή, γιατί γίνεται ευρεία χρήση αντιβιωτικών. Εμείς θα θέλαμε να συνεχίσουμε σε αυτή μας τη μάχη και θα υποστηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες προς αυτό το εγχείρημα. Υπ' αυτή την έννοια την 1η Μαρτίου του 2019 θα οργανώσουμε στο Βουκουρέστι μία υπουργική συνάντηση για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, όπου θα καλέσουμε τους Υπουργούς Υγείας από όλα τα κράτη-μέλη και εμπειρογνώμονες σε σχέση με την κτηνιατρική υγεία. Έτσι θα ορίσουμε τις κατάλληλες δράσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τα αποτελέσματα της διάσκεψης θα προτείνουμε ένα φάσμα συμπερασμάτων σε σχέση με αυτό το θέμα της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά. Και με βάση το One Health Approach η Προεδρία μας θα προβεί στον κατάλληλο συντονισμό για να φτάσουμε σε μια κοινή θέση σε σχέση με την μικροβιακή αντοχή στα αντιβιωτικά σε διεθνές επίπεδο. Σε σχέση με τον εμβολιασμό θα θέλαμε να συνεισφέρουμε με την, χρηστή, με την ανταλλαγή μάλλον χρηστών πρακτικών για μέτρα κάλυψης εμβολιακής ε, κάλυψης για τη δημόσια υγεία. Υπ' αυτή την έννοια στην Κλούς Λαπόκα, στην Τρανσιλβανία, θα γίνει ένα εργαστήρι για το πρόγραμμα εμβολιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη κάλυψη με βάση τις απειλές στη δημόσια υγεία. Θα καλέσουμε εμπειρογνώμονες και συντονιστές εθνικών προγραμμάτων και θα καλέσουμε και τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υγείας εξανατολών. Επίσης θα συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Μεταδοτικών Νόσων. Τα θέματα αυτά σχετίζονται με μια κοινή προσέγγιση των χωρών και των υποψηφίων επίσης χωρών για να ορίσουμε τα κοινά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αρθούν για να έχουμε τη βέλτιστη κάλυψη με βάση κοινή αγορά εμβολίων, κοινά προγράμματα και επίσης ε, θέματα που αφορούν τα αντιγόνα καθώς και την κατάσταση των μη εμβολιασμένων και τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν ως προς το μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμού. Σε σχέση με την πρόσβαση στα φάρμακα, η Προεδρία θα προωθήσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την πρόσβαση στα φάρμακα και στις ε, καινοτόμες θεραπείες σε λογικές τιμές, σε προσιτές τιμές για όλους και βελτίωση πρόσβασης έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή κάλυψη. Θα γίνει και μία άτυπη συνάντηση των Υπουργών Υγείας την 1η Απριλίου στο Φουκουρέστι. Κατά την άτυπη αυτή σύνοδο θα ασχοληθούμε και με την κινητικότητα των ασθενών μέσα στα πλαίσια της οδηγίας 204 του 2011 και για την διασυνοριακή κάλυψη υγείας. Θα δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, σπάνιες ασθένειες και ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους και την κάλυψη των σπανίων ασθενειών μέχρι τα 18 χρόνια. Επίσης, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες θεραπείες στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση σπανίων νόσων στις χώρες όπου προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη πολλές φορές γιατί πολλές φορές γίνεται χρήση γενώσιμων φαρμάκων και δεν έχουν πρόσβαση οι πάντες σε αυτά. Δυστυχώς δεν υπάρχει μία καλή διανομή γιατί πρόκειται για σπάνιες ασθένειες και οι, πολιτι... οι εθνικές πολιτικές δεν είναι πάντα οι ίδιες. Η ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας παράλληλα αποτελεί ένα θέμα ύψης της σημασίας και θα οργανώσουμε μια διυπουργική συνάντηση στα πλαίσια της e-health μαζί με το DigiConnect και τα Υπουργεία Τηλεπικοινωνιών. Θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε και τους ασθενείς οι οποίοι δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ασθένειες, ασθένειες με νεοπλασίες. Γι' αυτό θα οργανώσουμε στο Βουκουρέστι μια συνάντηση όπου θα καλέσουμε εμπειρογνώμονες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου. Δηλαδή, ιδιαίτερα ε, τον έλεγχο του καρκίνου, πρόληψη, θεραπεία και ευρωπαϊκές δράσεις καθώς και εθνικά προγράμματα στον τομέα της πρόληψης ε, και θεραπείας για να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την πρόληψη του καρκίνου. Αυτά είναι τα βασικότερα ε, προβλεπόμενα γεγονότα. 1η Μαρτίου στο Βουκουρέστι, Υπουργική Συνάντηση για τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ε, μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά και στη συνέχεια θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα συμπερασμάτων. Στις 21-22 Μαρτίου στο Βουκουρέστι θα γίνει η συνάντηση των επικεφαλής ε, των τμήματων ιατρικής πρόληψης για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το θέμα οι ειδικοί. Στη συνέχεια, η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Υγείας στις 14-15 Απριλίου, όπου θα θίξουμε θέματα όπως την καθολική πρόσβαση στα ε, φάρμακα, αντιμετώπιση της υπατήτηδας γάμα και εφαρμογή της οδηγίας 204 ε, του 2011, επτά χρόνια μετά την εφαρμογή της. Στις 9-10 ε, Μαΐου στην Κλούς ε, Ναπόκα θα γίνει μια συνάντηση για τον εμβολιασμό και την κάλυψη του πληθυσμού για θέματα δημόσιας υγείας και στις 4 Ιουνίου θα γίνει η συνάντηση ομάδας εργασίας, ένα σεμινάριο δηλαδή, σε επίπεδο κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την πρόληψη και την ανείχνευση του καρκίνου στα πρώιμα στάδια. Και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουμε την ψηφιακή υγεία σε μια συνάντηση του Ιουνίου του 2019. Η θητεία μας ε, στην ουσία θα καλύψει και θέματα ύψης της σημασίας όπως το Brexit, τις ευρωεκλογές και τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύουμε όμως ότι θα έχουμε μία φιλόδοξη εντολή καλύπτοντας τις ε, ανάγκες των πολιτών και θα θέλαμε και εσείς και γνωρίζουμε ότι εσείς είσαστε ένας σημαντικός μας εταίρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό για αυτή την παρουσίαση. Και φυσικά θα έχουμε και ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Συνάδελφοι, ο συνήθως θα γίνει ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους τους. Δύο λεπτά ο καθένας. Μετά θα απαντήσει η υπουργό και θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος ερωτήσεων για τα μέλη με χρόνο αγόρευσης ενός λεπτού. Ποιος Μπέλετ έχει το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας καλωσορίζω θερμά κυρία Υπουργέ. Καλή χρονιά, καλή επιτυχία στη Ρουμανική Προεδρία. Είπατε ότι είσαστε πολύ φιλόδοξοι. Μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Νομίζω ότι συμφωνούμε με όλες αυτές τις προτεραιότητες. Τις συμμεριζόμαστε. Και σίγουρα θα σας στηρίξουμε. Είπατε ότι όλοι εργαζόμαστε προς όφελος των πολιτών και των ασθενών. Η κυρία Βαλεάν είπε ότι οι δικές σα αρμοδιότητες είναι εξαιρετικά σημαντικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα για την Επιτροπή μας. Δύο θέματα θέλω να θίξω ιδιαίτερω. Πρώτον, οι, προτεραιότητε σα είναι και δικές μας προτεραιότητες, αλλά τι γίνεται με τα λεφτά, με τον προπολογισμό. Στο τρέχον στο δημοσιονομικό πλαίσιο γνωρίζουμε τι έχουμε διαθέσιμο. Τι όμως θα γίνει στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2021. Προφανώς οι συζητήσει δεν θα ολοκληρωθούν πριν το καλοκαίρι, αλλά εσείς ε, παίζετε σημαντικό ρόλο, οπότε είστε πρόθυμοι να στηρίξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα όσα ζητάει για ε, ένα αυτόνομο, πλήρω αυτόνομο πρόγραμμα υγεία για την επόμενη προγραμματική περίοδο σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή, θα καλωσορίζαμε την υποστήριξή σας. Δεύτερον, η κινητικότητα των ασθενών είναι μία από τις προτεραιότητές σας. Το στηρίζουμε. Είμαι συμπτωματικά εισηγητή στην έκθεση για την εφαρμογή της ε, οδηγίας υπηρεσιών διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας και μπορώ να σας πω ότι ε, η εισήγησή μου, η γνωμή μου έλαβε μεγάλη πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή. Την επόμενη μήνα θα πάει στην Ολομέλεια. Ε, μιλήσατε για τις ε, χρόνιες ασθένειες, σπάνιες ασθένειες που χρειάζονται ιδιαίτερες θεραπείες. Ένα από τα στοιχεία τα οποία συζητήσαμε το πρωί είναι το αίτημα σε εσά και στην Κομισιόν να, το, το αίτημα να δημιουργηθούν όχι να δημιουργηθούν καινούργια κέντρα, αλλά κέντρα που υπάρχουν ήδη να εξειδικευθούν, νοσοκομεία συγκεκριμένα κλπ, να εξειδικευθούν σε χρόνιες ασθένειες, ε, θεραπεία του καρκίνου, συγκεκριμένα ειδικά, δηλαδή θέματα ειδικέ παθολογίες, για τις οποίες θα στηρίζαμε αυτά τα κέντρα να ειδικευθούν έτσι ώστε να στηρίξουν μετά και την κινητικότητα των ασθενών. Ευχαριστώ. Uh, Κυρία Σέρμπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο το θέμα που θα, που θα ήθελα μάλλον να θίξω είναι η πολυσαρκία. Η προτεραιότητα της Μάλτας έθιξε το θέμα της, πολυσ... παχυσαρκίας, με συγχωρείτε, και ιδιαίτερα της παχυσαρκίας των ανηλίκων, των μικρών παιδιών. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα η Ρουμανική Προεδρία και δεν, δεν ξέρω κατά πόσο προβλέπετε ένα νέο πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Ο κύριος Πιέκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω θερμότατα στη σημερινή μας συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ. Παρουσιάσατε εκτενώς τις προτεραιότητες της ε, Ρουμανικής Προεδρίας και το πρόγραμμά σας για το ερχόμενο εξάμεινο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με τα τρέχοντα ζητήματα, τα νομοθετικά που είναι πάντα δύσκολα και ένα δεύτερο ερώτημα για το μέλλον. Για τα τρέχοντα νομοθετικά ζητήματα, το Δεκέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση ε, για την έκθεση αξιολόγησης των τεχνολογιών των ιατρικών. Στόχο έχει αυτή ε, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και ε, οι διπλοδουλειές εμπολής για το ίδιο θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή της Κομισιόν την ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν από τρεις μήνες περίπου. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξη αυτή η πρόταση. Εξ όσων γνωρίζω, το Συμβούλιο δεν έχει κατενθουσιαστεί με την συγκεκριμένη εκθέση. Και ρωτώ, κυρία Υπουργέ, εσείς πώς το βλέπετε. Πιστεύετε ότι το επόμενο εξάμεινο μπορεί κάτι να γίνει, να βρεθεί κάποια συνένεση για το συγκεκριμένο θέμα στο Συμβούλιο. Γιατί είναι και νομοθετικού περιεχομένου η έκθεση για την αξιολόγηση των ιατρικών τεχνολογιών, των τεχνολογικών υγείας. Και ένα άλλο ερώτημα λίγο πιο απότερο. Στην ιατρική υπάρχει το θέμα της τεχνητής της νοημοσύνης. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό κάπως φουτουριστικό, επιστημονική φαντασία, αλλά γνωρίζουμε ότι ήδη ε, στα νοσοκομεία υπάρχουν μηχανήματα ε, που αναλαμβάνουν κάποιες βοηθητικές ε, λειτουργίες ε, με υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ρουμανική Προεδρία προτίθεται να ε, προωθήσει ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική. Δεν είναι ευκαταφρόνητο αυτό το θέμα, γιατί η τεχνολογική πρόοδος καλπάζει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς τώρα να αφυπνιστούμε και να ασχοληθούμε και με τις νομικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρία Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Ε, σας εύχομαι ειλικρινά επιτυχία για την πρώτη σας Προεδρία. Ε, Είπατε σύντομα ότι έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υγεία με κάποιε προτεραιότητε. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω σε ορισμένε. Μιλήσατε πολύ για την αντίσταση των ε, μικροβίων στα αντιβιωτικά. Εδώ και καιρό αποτελεί αυτή η προτεραιότητα στα θέματα υγεία στην Ευρώπη. Είναι πολλοί εμπειρογνώμονε που θεωρούν ότι αυτή μπορεί να γίνει απειλή ε, πιο σημαντική από τον ίδιο τον καρκίνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πέρσι τον Οκτώβριο το Κοινοβούλιο μα ενέκρινε την έκθεση Κάντενμπαχ με ένα ψήφισμα πάρα πολύ στεναρό προς την κατεύθυνση αυτή και ε, αντανακλά και κάποια αριθμητικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δήλωση και Ελέγχου Νοσημάτων. 4 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη όταν νοσηλεύονται ε, ε, προσβάλλονται από ενδονοσοκομιακές νόσους και 37.000 χάνουν τη ζωή τους ως συνέπεια. Εσείς λοιπόν πώς θέλετε να προχωρήσετε. Ξέρω ότι έχει αρχίσει η συζήτηση για την ευαισθητοποίηση ε, και των ασθενών και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά πέρα από αυτό να μην μειώσουμε κάποια στιγμή τη χρήση των αντιβιωτικών. Και μάλιστα ε, να έχουμε και μια πολιτική τιμολογιακή που να αποθαρρύνει, να ενθαρρύνει. Θέλω να μιλήσω για την όσο του Λάιμ τώρα επίσης τηλεγραφικά. 800.000 ε, είναι οι Ευρωπαίοι που υποφέρουν από την όσο αυτή και εκεί το Κοινοβούλιο προχώρησε. Η δική σας Προεδρία έχει την πρόθεση να το θέσει αυτό το θέμα επιτάπητος και να εγκρίνεται ένα πρόγραμμα δράσης με συστάσεις για το Συμβούλιο. Και ένα τελευταίο, έχετε όλη την υποστήριξή μας ε, για το θέμα των σπανίων νόσων, στο οποίο αναφερθήκατε, εχθές με κάποιους εμπειρογνώμονες ε, και κάποια ε, σωματεία και ενώσεις λανσάραμε ένα πρόγραμμα για το 2030, μέχρι το 2030 είναι στη διάθεσή σας για να προχωρήσετε, για να σας υποστηρίξουν για να προτείνετε πολιτικές που να απαντούν σε αυτές τις αρρώστιες μπορεί να είναι σπάνιες αρρώστιες είναι 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, καλώς ορίσατε εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ εξελέγη το 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και είπα και στον πρόεδρο Ιωάννης και στους Ρουμάνους βουλευτές και σε άλλους ε, και τους ρωτούσα άλλο και περισσότερο τι γίνεται με τα δέσποτα σκυλιά στους δρόμους σας. Και είναι πονίδιστο αυτό που έζησα. Δεν μου απαντούσαν ή ε, απέφευγαν να μου απαντήσουν γιατί είναι ε, πραγματικά τεράστια τα δεινά στα οποία υποβάλλονται αυτά τα δέσποτα ζώα. Εσείς επιτέλους μπορείτε να μου απαντήσετε ήδη από το 2014 εδώ στο Κοινοβούλιο Ε, ε, ε, δώσαμε μια επιστολή ε, ένα χαρτί το οποίο κάλυπτε απόσταση ενός χιλιόμετρου από μαθητές και πάρα πολλοί μαθητές ήταν από τη Ρουμανία. Ήταν παιδιά που είχαν ζήσει τεράστιες ε, ψυχικά τραύματα. Εγώ πήρα εκατοντάδες email και γράμματα από παιδιά από τη Ρουμανία και πραγματικά μου σπάραξε η καρδιά διαβάζοντας αυτά τα γράμματα. Εσείς κυρία Επίτροπε, τι προτίθεστε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτά τα ψυχικά τραύματα, αυτά που ζουν οι Ρουμάνοι και ιδιαίτερα τα παιδιά στη Ρουμανία βλέπουν με πιο φρικτό τρόπο φέρεται ο κόσμος στα δέσποτα σκυλιά. Το ζουν στο πετσί τους. Και είναι υποχρεωμένα να υφίστανται αυτέ τι εικόνε και αυτά τα τραύματα. Δεύτερον, επειδή τα δέσποτα σκυλιά ε, γενικά δεν ε, εμβολιάζονται κατά τη λύσα και δεν έχουν και μικροτσίπ. Και είναι και πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των Ρουμάνων πολιτών. Εκεί τι προτίθεστε εσεί να κάνετε. Και μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο η χώρα σα δεν διώκει ε, αυτή την κατάσταση και δεν το διαχειρίζεται. Οι περισσότεροι στην Ευρώπη καταδικάζουν αυτή την εικόνα στη χώρα σας και πλήττεται και το κύρο στη Ρουμανία. Πέρα από τα άλλα αρνητικά που δεν θέλω τώρα να αναφέρω, πλήττεται πάρα πολύ σφοδρά. Ε, ε, αδιαφορεί τελείω η ρουμανική κυβέρνηση για το τι σκέφτονται άλλοι πολίτες για τη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη κύριε Εκάουτ, δική σας ήταν η σειρά. Σας καθυστερήσαμε λίγο, έχετε τώρα το λόγο. Κανένα πρόβλημα, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την εισαγωγή σας, για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας. Και όταν μιλάμε για την κινητικότητα των ασθενών και τις σπάνιες ασθένειες, είναι οι προτεραιότητες τις οποίες τις μοιράζεται μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένω να ακούσω την απάντησή σας και στον κύριο Μπελέτ για πράγματα τα οποία εμείς συζητήσαμε επ' ευκαιρία της επεξεργασίας της νομοδότησης για τις σπάνιες ασθένειες, για τις και των ασθενών, συγγνώμη. Ε, δύο ακόμα πράγματα έχω να σας πω. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε την υγεία ως προτεραιότητά της. Ε, ήταν, ε, η αντίδραση ήταν πολύ αργή σε σχέση με πολλά θέματα τα οποία άπτονται τη υγείας. Είναι σημαντικό όμως οι προεδρίες να δίνουν βάρος σε αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε εσεί στα εξή δύο. Αντιμικροβιακή αντίσταση, την οποία ανέφερε και η συνάδελφο κυρία Ρή. Ξέρουμε ότι το 2017 η Κομισιόν είχε υποβάλει ένα πρόγραμμα δράσης για την ε, κατά τη αντοχής στα αντιβιωτικά. Και ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του πράγματος ήταν ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να γίνει ε, περιοχή βέλτιστων πρακτικών, ζώνη βέλτιστων πρακτικών. Συχνά βέβαια το λέμε αυτό χωρίς να συμβαίνει τίποτα τελικά. Πώς λοιπόν σκοπεύει η Ρουμανική Προεδρία να προωθήσει τη συζήτηση αυτού του θέματος και στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη έτσι ώστε πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί μια περιοχή βέλτιστων πρακτικών για το θέμα των, ε, της αντιμικροιακής αντίστασης. Ε, επίσης, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Η Κομισιόν και για αυτό το θέμα έχει υποβάλει μια ανακοίνωση τον περασμένο Νοέμβρη. Εμεί στο 7ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον είχαμε πει ότι το 2018, πέρσι δηλαδή, θα έπρεπε να έχουμε διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση στην έκθεση σε ενδοκρινικού διαταράκτε. Συνεπώ, έχουμε στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Το συμφωνήσαμε αυτό στο 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράση. Από τότε από την Κομισιόν καμία αντίδραση. Οπότε περιμένουμε από την Προεδρία, τη Ρουμανική Προεδρία, να δώσει έμφαση και σε αυτό το θέμα, θέμα έτσι ώστε στην Ευρώπη πράγματι να εξασφαλίσουμε ένα μη τοξικό περιβάλλον. like this when have a presidency invited, so you have to commit and. Uh, ε, τώρα να δώσω το λόγο στην Υπουργό για να μας πει ε, πώς θεωρεί η Ρουμανική Προεδρία ότι πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα σε σχέση με αυτά που έκανε ή δεν έκανε η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω τι θα κάνει η Ρουμανία, λέει η Υπουργός Υγείας. Θα αρχίσω με, τον, με το ερώτημα του κυρίου Μπέλετ. Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας και χαίρομαι για τις προτεραιότητες που έχετε και εσείς και εμείς. Και βλέπω ότι κατά ένα μεγάλο μέρος συμπίπτουν. Κύριε Μπέλετ, θα αρχίσω με τη δεύτερη ερώτηση Όταν συζητήσαμε για τους στόχους της Ρουμανίας μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας, είχαμε κατά νου την ίση πρόσβαση στην υγεία όλων των πολιτών. Και επειδή συναντήθηκα και συνάντησα πολλαπλά προβλήματα για ε, την αντιμετώπιση των σπανίων παθήσεων και μετά από την εξέταση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και συζητώντας τα αποτελέσματά της καθώς και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι έμπρακτα. Μιλήσατε για αυτά τα κέντρα αριστείας ε, για την αντιμετώπιση των ε, σπανίων ασθενειών. Ε, ένιωσα ότι υπήρξε απόλυτη σύμπτωση απόψεων, διότι αυτό με είχε απασχολήσει ιδιαίτερα και στη Ρουμανία. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε τους ασθενείς αυτούς ενδοευρωπαϊκά. Σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα υποστηρίξω την Επιτροπή για την καλύτερη κατανομή των πόρων για την κάλυψη των αναγκών υγείας και πιστεύω ότι και εσείς ε, θα κάνετε το ίδιο γιατί η υγεία πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όλοι οι πολίτες ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγεία ισότιμα. Ως προς το ερώτημα της ε, κυρίας Σέρμπου, θα ήθελα καταρχήν να σας ε, συγχαρώ για θέματα που σας απασχόλησαν σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και την αντιμετώπιση του θέματος της παιδικής παχυσαρκίας. Έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα ως Ευρωβουλευτής αλλά και ως μητέρα. Το θέμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας είναι κάτι το οποίο μας απασχόλησε, θα δοθεί τελική μορφή σε αυτό το σχέδιο το 2019, αλλά στην ατζέντα μας δεν έχει ενταχθεί αυτός ο στόχος, όμως θα συνεργαστώ με τη Φιλανδική Επικείμενη Προεδρία επί του θέματος. Θα ήθελα να σας ε, μιλήσω και για καλά νέα από τη Ρουμανία, γιατί χτες δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα ο νέος νόμος για την εκπαίδευση, ε, βάσει του οποίου οι Υπουργοί Εκπαίδευσης και Υγείας θα καταρτήσουν μια στρατηγική για την υγεία και την διατροφή για το σχολικό έτος. Άρα θα προωθήσουμε αυτή την στρατηγική και το πρόγραμμα στα σχολεία και είμαι σίγουρη ότι θα μας συνοδεύσετε σε αυτή μας την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με την τεχνολογική αποτίμηση της υγείας, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση την πρόταση κανονισμού. Αυτό είναι ένα από τα πέντε θέματα προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας γιατί και οι ασθενείς και τα προγράμματα υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τις τεχνολογίες εχμής. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια των ομάδων εργασίας εμπειρογνωμών στο Συμβούλιο. Παράλληλα, θα σας μιλήσουμε για, ε, για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, στο, που θα επιτελεστεί ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας ε, τον Ιούνιο στο Λουξεμβούργο. Ε, το θέμα είναι και θέμα χρόνου. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2018 εκκίνησε αυτό το πρόγραμμα. Χρειάζεται όμως περισσότερος χρόνος. Γι' αυτό και σας είπα ότι θα ήθελα να γίνει πρόοδος, άμεσα θα κάνω και διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους μου έτσι ώστε να γίνει έμπρακτα πρόοδος. Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, Είδατε στην παρουσίασή μου ότι ένα από τα θέματα άμεσης προτεραιότητας είναι το e-health, η ψηφιακή υγεία και πιστεύω ότι αυτά τα θέματα θα τα θίξουμε κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εβδομάδας 12 με 15 Ιουνίου μαζί με τον Υπουργό τηλεπικοινωνιών. Αλλά θα προωθήσουμε φυσικά και την δική σας ιδέα μέσα στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης. Προς την κυρία Ρης, θα ήθελα να πω τα εξής. Μιλήσαμε ακριβώς για αυτό το ε, θέμα της ε, μικροβιακής αντίστασης στα αντιβιωτικά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πρώτες 10 απειλές κατά της δημόσιας υγείας και φυσικά η μικροβιακή αντίσταση ήταν ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και μας απασχολούν. Είναι, ένα, είναι μία από τις βασικές απειλές κατά της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό προωθούμε και το θέμα του εμβολιασμού. Με το εμβόλιο κατά της γρήψης αλλά και άλλα εμβόλια. Την 1η ε, Μαρτίου του 19 θα οργανώσουμε μία διάσκεψη στο Βουκουρέστι για τα επόμενα βήματα ως ε, προς τις ε, βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντίστασης. Θα καλέσουμε τους Υπουργούς Υγείας από το κράτη-μέλη και θα φτάσουμε και σε ορισμένα συμπεράσματα σε σχέση ακριβώς με τις νοσοκομιακές λοιμώξεις και την μικροβιακή αντίσταση στα αντιβιωτικά. Μιλάμε για θέματα υγείας, περιβάλλοντος, γεωργίας. Έχουμε βεβαίως εστιάσει την προσοχή μας σε θέματα υγείας λόγω χαρτοφυλακίου, αλλά θα θέλαμε να γίνει, να γίνει μια συζήτηση και για τις λοιμώξεις στα νοσοκομεία. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δράσης, όπως είπατε και εσείς, για να μην παραμείνουμε σε ασκήσεις επί χάρτου. Γιατί Σύμφωνα, με τα νέα στατιστικά στοιχεία, οι νοσοκομιακές λοιμώξεις έχουν πολλαπλασιαστεί ανησυχητικά. Σε σχέση με την νόσο του ΛΑΙΜ. Η πρόταση νομοθετική, νομοθετικού περιεχομένου είναι ένα θέμα αρμοδιότητας της Κομισιόν. Μετά το Συμβούλιο θα αποφανθεί. Ο κύριος Εκ υπέβαλε επίσης ένα ερώτημα σε σχέση με τα αδέσποτα σκυλιά που δεν έχουν ενταχθεί στη βασική μας ατζέντα, ξέρω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις επί του θέματος. Έχω, μια προσωπική, έχω προσωπική γνώμη επί του θέματος. Ξέρετε ότι ίσως δεν ξέρετε, ότι εγώ έχω υιοθετήσει τρεις ε, αδέσποτες γάτες και δύο σκυλιά. Αυτό υπό προσωπικού επίπεδου. Τώρα, σε σχέση με το έτος ε, μικροβιακής αντίστασης, έχετε απόλυτο δίκιο. Το 2017 οι χώρες ενέκριναν ένα πρόγραμμα δράσεις για την ε, μικροβιακή αντίσταση στα αντιβιωτικά. Θεωρήσαμε ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να ενταχθεί για να βρούμε συγκεκριμένες ε, και σφαιρικές λύσεις. Ε, θα ήθελα να σας πω τι κάνει η Ρουμανία αυτή τη στιγμή. Πέρσι τον Οκτώβριο η κυβέρνηση αποφάσισε να προβεί σύσταση μιας διυπουργικής επιτροπής ακριβώς για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Συμμετείχαν και συμμετέχουν εμπειρογνώμενες από όλα τα Υπουργεία και προβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις. Όμως, πέρα από αυτό, το πρώτο βασικό βήμα ήταν το θέμα της αναγνώρισης για να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα έχουμε κάνει μέχρι τούδε. Ε, παραμένουμε ανοιχτοί σε προτάσεις, θα σας ε, προβάλλουμε, θα σας αναφέρουμε τα συμπεράσματα της ε, διάσκεψης του Μαρτίου και θα θέλαμε να πλαισιώσετε τις δράσεις μας για να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα και για να έχουμε και σημαντικούς δείκτες, θετικούς δείκτες. Ως προς το το δεύτερο θέμα που θίξατε, δηλαδή για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες, περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής. Αυτά μπορώ να σας πω μέχρι τώρα. Ωραία, τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο. Ο καθένας έχει ένα λεπτό για να υποβάλει την ερώτησή του. Ο, κύριος ο, ο πρώτος είναι ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, κυρία Υπουργέ. Συμφωνώ και εγώ με τον Ιβο Μπέλετ. Έχει μεγάλη σημασία το μελλοντικό πρόγραμμα υγείας με βάση τις διαπραγματεύσεις και την αύξηση του προϋπολογισμού για να φτάσουμε σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την υγεία, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα Χαίρομαι γιατί μία από τις προτεραιότητες είναι ο εμβολιασμό. Υπάρχει αύξηση των ε, νόσων στη Ρουμανία αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πώς θα υπάρχει μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας μεταξύ κρατών για τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού ως προς τις ε, νέες τεχνολογίες στον τομέα της ιατρικής, θα ήθελα να υπάρξει μια γενική συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και να ε, δημιουργηθούν αυτά τα τρία περιφερειακά νοσοκομεία στη Ρουμανία, να ε, συσταθούν αυτά τα νοσοκομεία για να μην χάσουμε και τα χρήματα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καβεσόν Ρουίς. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για όσα μας είπατε. Να πω κατευθείαν στο ψητό για την αξιολόγηση των ε, τεχνολογιών υγείας. Φιλόδοξο το, φιλόδοξη αυτή η προτεραιότητα, ε, παρόλο ότι περιμένουμε την ε, Κομισιόν μέχρι τον Ιούνιο. Ε, οπότε ίσως μετά το τέλος θητείας μας. Το σημαντικό όμως είναι το Συμβούλιο να είναι όσο πιο επικοδηματικό γίνεται. Η πρόταση της, ε, του Κοινοβουλίου ε, ήταν παρόμοια αυτή του Συμβουλίου τώρα. Οπότε ο διάλογος καλό θα είναι να γίνει επικοδομητικός χωρίς μπλοκαρίσματα. Να μην συνεχίζουμε να παραπονιόμαστε για την πρόσβαση στα φάρμακα και το Συμβούλιο να μην κάνει τίποτα. Μετά, ε, η έλλειψη ε, φαρμάκων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον. Στο Κοινοβούλιο αύριο ψηφίζεται ένα σχετικό κείμενο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει ε, να βγει στην αγορά κυταρικές θεραπείες. Ε, χρειάζεται να τις μελετήσουμε και ομοιοπαθική. Να, να, να ξαναδούμε λίγο την οδηγία γιατί τα ομοιοπαθικά δεν είναι φάρμακα, ε, δεν έχουν εγκριθεί ως τέτοια, παρόλα αυτά αποκαλούνται φάρμακα. Μετά, η πατήτιδα C, C ε, πατήτα Γ χρειάζεται ένα σχέδιο εκρίζωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιέκα. ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε. Όλοι μίλησαν εδώ ε, για την ε, αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Το είδαμε αυτό από την Ολλανδική Προεδρία. Και σήμερα το πρωί το συζητήσαμε και με τον άλλο Υπουργό ε, γεωργίας ε, και θα γίνει και μια διάσκεψη και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ε, να συμμετέχουν και ευρωβουλευτές που είναι ειδικοί και αλληλεμπειρογνώμονες. Καλό είναι να καλείτε υπουργού, αλλά πρέπει να καλείτε και εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. είμαστε συμπληρωματικοί στη δράση μας και γνωρίζουμε και εμεί πράγματα. Και διακομματικό αυτό δεν έχει να κάνει με παρατάξει. Και τέλος ε, οι προληπτικοί εμβολιασμοί ε, στα νεογνά είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνετε με μέτρα έτσι ώστε και οι σύγχρονοι γονείς να μην σκέφτονται ότι καλά δεν χρειάζεται να το εμβολιάσω το μωρό μου τώρα και μετά αυξάνονται οι ασθένειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Παχνιού. Όπω Όπως το είπατε και εσείς και το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, στην καρδιάρκεια τη της σας ε, έχετε προτεραιότητα στην πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα για ε, παιδιά με βαριές ασθένειες. Σήμερα η φαρμακοβιομηχανία καθορίζει την τιμή αυτών των φαρμάκων ε, σε συνάρτηση με τις με το στάτους της αγοράς. Ε, ένα φάρμακο για την πατήτα γάμα, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίσει 49.000 ευρώ στις ΗΠΑ, 41.000 στη Γαλλία, 4.000 στην Ταϊλάνδη και 700 στην Αίγυπτο. Το ίδιο ακριβώς φάρμακο. Για να λήξουν αυτές τις πρακτικές χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα λαμβάνει υπόψη ότι τα καινοτόμα φάρμακα δεν είναι καταναλωτικά αγαθά όπως όλα τα υπόλοιπα, αλλά που η χρήση τους είναι ανάγκη και όχι επιλογή. Οπότε θέλετε να ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο της καινούριας οδηγίας για την διαφάνεια στον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν έχει αποσύρει την αρχική της νομοθετική πρόταση το Δεκέμβριο του 2000. 2014. Ε, ε, δεν θα έπρεπε όμως να ξαναζητήσει πρόταση το Συμβούλιο γι' αυτό, νομοθετική πρόταση του για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Thank you too, Mr. Now, Mr. Zani. Κύριο Ζάνι. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω να κάνω. αφού συμφωνήσω με όσους μίλησαν προηγουμένως για τις ευάλωτε ομάδες του πληθυσμού μας και κυρίως τα παιδιά. Και δεν μιλώ μόνο για, τη, τα εμβόλια ή τις μεταδοτικές ασθένειες που είναι σίγουρα πολύ σημαντικά θέματα. Μιλώ για την πρόσβαση στα φάρμακα. Για παιδιά, για παράδειγμα, που ε, έχουν διαβήτη όλο και περισσότερα. Με εκθετικό βαθμό αυξάνονται αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο για τις οικογένειές τους να βρουν τα ποσά που χρειάζονται για να ε, τα πάρουν τα παιδιά τους. Πρόκειται για φάρμακα που είναι σχετικά ακριβά. Επίσης έχουμε ε, την παχυσαρκία, ένα άλλο θέμα για το οποίο χρειάζεται μια εκστρατεία ενημέρωση του πληθυσμού. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Ρουμανική Προεδρία σκοπεύει να κάνει κάτι και για τους ε, πιο ηλικιωμένου και για την πρόσβασή τους στα φάρμακα. Για παράδειγμα φάρμακα μείωση της πίεσης. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ε, ατόμων πεθαίνουν από αυτά τα αίτια γιατί δεν έχουν πρόσβαση για οικονομικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούτλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, κυρία Υπουργέ. Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά τα έχετε στο κέντρο της μέρημνάς σας. Είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας κλπ. Δύο ερωτήσεις για αυτό το θέμα των παιδιών. Πρώτον, ε, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Περιμένετε, είπατε, η Κομισιόν να υποβάλει το πρόγραμμα δράσης που ετοιμάζει. Πόσο θα περιμένουμε, δεδομένου ότι η Κομισιόν στο παρελθόν για αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι, ήταν πολύ αργή. Πώς ε, θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία απαλλαγμένη από υψηλού κινδύνου ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα. Υπάρχουν μελέτες που συνδέουν τις ορμόνες στα παιδιά και τις μελλοντικέ ασθένειες από τις οποίες θα πάσχουν. Θα ήθελα η Ρουμανική Προεδρία να ηγηθεί της προσπάθειας να δείξει αποφασιστικότητα. Χρειαζόμαστε μια οριζόντια νομοθεσία που θα προστατεύει πραγματικά και συνολικά τον πληθυσμό. Θέλουμε το πρόβλημα αυτό να λυθεί οριζοντίως. Ερώτηση λοιπόν θα ταρακουνήσει λίγο την Κομισιόν το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Δεύτερον, και πάλι για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν παντού την ίδια πρόσβαση στα φάρμακα της θεραπείας. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Κύριο Στανασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη μικρή μας οικογένεια που είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί το θέμα του εμβολιασμού, των εμβολιασμών, είναι ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γιατί η Ρουμανία είναι μία από τις χώρες όπου είδαμε μία αναζωπήρωση συγκεκριμένων νόσων που θεωρούσαμε ότι βρίσκονται κοντά στην εξάλληψη, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και διότι αυτό ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το τελευταίο καιρό. Και άλλοι συνάδελφοι ανησυχούν για αυτές τις εξελίξεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Όπως είπατε, μία από τις προτεραιότητες σας είναι οι εμβολιασμοί. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, τελευταία σύσταση του Συμβουλίου για, την, ε, για το εύρος της κάλυψης, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προβλέπει η Ρουμανική Προεδρία να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα που προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ήταν και ο δεύτερος ε, γύρος, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Έχετε το λόγο, κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Κριστιαν Μπουσόη καταρχήν ε, με βάση την τελευταία του ερώτηση. Φυσικά θα προβούμε στην οικοδόμηση των τριών περιφερειακών νοσοκομείων στη Ρουμανία και θα γίνει αυτό με ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν θα χάσουμε αυτά τα χρήματα και αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το άνοιγμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ως προς το πρώτο ερώτημα σε σχέση με τους εμβολιασμού, πράγματι οι εμβολιασμοί είναι ένα από τα θέματα που προωθεί η Ρουμανική Προεδρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό, όπως σας είπα ήδη, στην κλουσνα Πόκα το Μάιο θα οργανωθεί ένα εργαστήριο για τα προγράμματα εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μεγαλύτερη κάλυψη του πληθυσμού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για άλλη μία φορά τις πρώτες 10, ότι μέσα στις πρώτες 10 προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών είναι και το θέμα της ευρύτερης κάλυψης του πληθυσμού ως προς τους εμβολιασμούς. Θα θέλαμε λοιπόν μαζί με τους εμπειρογνώμενες που θα καλέσουμε σε αυτή τη ε, διάσκεψη να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις ε, για να καταδείξουμε τι συμβαίνει εμβολιασμός. Θα προβούμε σε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και θα ε, ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε μια στρατηγική και ειδικά μέτρα για την αύξηση της ε, κάλυψης των εμβολιασμών ως προς τη μετανάστευση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό εμβολιασμών για να δούμε ποιο είναι το εύρος της κάλυψης και θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Τανασέσκου το εξής. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα προσκόμματα που υπάρχουν, τα κοινά εμπόδια ως προς την μεγαλύτερη εμβολιακή κάλυψη. Και θα πρέπει να εφαρμόσουμε και τις βέλτιστες πρακτικές που έδωσαν αυτά αποτελέσματα στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μιλήσω και για μία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ρουμανία. Πέρσι το Μάιο, μαζί με ε, εμπειρογνώμονες της UNICEF και του ΠΟΗ, άρχισε μία ε, πρωτοβουλία πόρτα-πόρτα δηλαδή για τους πολίτες που δεν είχαν πρόσβαση σε, στις ιατρικές υπηρεσίες, που δεν είχαν τον οικογενειακό τους γιατρό. Γιατί είχαμε πολλά κρούσματα ηλαράς πέρσι στη Ρουμανία. Προσπαθήσαμε να βρούμε μία λύση, να βρούμε εμβόλια χωρίς αποτέλεσμα χωρίς σοβαρά αποτελέσματα. Ήταν μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία που εντάχθηκε και στην ατζέντα της UNICEF. Και μπορώ να σας πω ότι σε μια κοινότητα που είχε κάλυψη 3,9% κάλυψη εμβολιασμού φτάσαμε σχεδόν στο 100% κάλυψης με την βοήθεια επιδημιολόγων, γιατρών κλπ. Ελπίζω και στην Κλούσνα Πόκα να φτάσουμε σε πολύ καλά αποτελέσματα και πρακτικές για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο ε, υπ' αυτή την έννοια. Σας μίλησα και για τον ΠΟΗ γιατί με βάση την αύξηση κάλυψης κατά 10% θα σώσουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό, κάτι που επιθυμούμε όλοι και που είναι ένα αποτέλεσμα ουσίας σε σχέση με την ε, τεχνολογική αποτίμηση υγείας, όπως σας είπα κύριε Μπουσόη, η Ρουμανία θα ήθελε να έχει ουσιαστική πρόοδο. Ο στόχος μας βεβαίως είναι πολύ φιλόδοξος γιατί πολεμάμε με το χρόνο και για να υπάρξει ε, ένα κανονιστικό πλαίσιο και μία εναρμόνιση χρειάζεται χρόνος, αλλά θα καταβάλουμε προσπάθειες και θα γίνουν και διμερείς συναντήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο ως προτεραιότητα ως προς την στρατηγική επικοινωνία υπέρ του εμβολιασμού. Βεβαίως είναι ένα θέμα εθνικής αρμοδιότητας και θα πρέπει να προωθηθεί σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Αλλά θα υπάρχει και μία κοινή προσέγγιση. Ο Υπουργός Ντάεα σας μίλησε για τη διάσκεψη της 1ης Μαρτίου για την αντίσταση στα αντιβιωτικά και σας είπα ότι φυσικά ε, υπάρχουν και νοσοκομιακές λοιμώξεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να δούμε τι επικρατεί και στον αγροτικό κόσμο, τι επικρατεί στην Ήπεθρο. Γι' αυτό θα ήθελα να έρθετε σε αυτή τη διάσκεψη, γιατί νομίζω ότι θα συζητηθούν πολλά και θα φτάσουμε και συγκεκριμένα συμπεράσματα, πιστεύω. Άρα σας καλώ επίσημα στη διάσκεψη αυτή του Μαρτίου. Νομίζω ότι το ίδιο έκανε και ο Υπουργός Ντάε το πρωί. Θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Παρνιέ. Παρνιό. Εμείς ε, θέλουμε να προβάλλουμε και πρωτοβουλίες στο θέμα της διαφάνειας και πρόσβαση στα φαρμακευτικά σκευάσματα. Και θα ήθελα να πω το εξή. Στη Ρουμανία έχουμε κάνει σημαντικά ε, βήματα για την αντιμετώπιση της υπατήτηδας γάμα. Μπορώ να σας πω ως Υπουργός Υγείας ότι υπάρχουν ε, τα ε, λεγόμενα προγράμματα ε, αντιμετώπισης ασθένειας της, της πνευμονικής πνευμονο Σύνοσης με Ιντερφερόνι. Μιλάμε για την πρόσβαση των ασθενών στην υγεία και στα φαρμακευτικά σκευάσματα. Στις 14-15 Απριλίου θα γίνει μια σύσκεψη στο Βουκουρέστι και είμαι πεπισμένη ότι θα γίνει λόγος ε, για την καθολική πρόσβαση στα φάρμακα. Όταν μιλάμε για ε, παιδιά και γενικά ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει να υπάρχει καθολική πρόσβαση στα πράγματα, ε, στα, προγράμματα υγείας. Έχουμε και ένα εθνικό πρόγραμμα στη Ρουμανία, το οποίο επεκτάθηκε πέρσι, για να υπάρχει και ένα πρόγραμμα ελέγχου των παιδιών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Άρα θα το δούμε και αυτό το θέμα πανευρωπαϊκά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το υπενθυμίσατε. pentru doamna deputat Guteland. Ως προς ε, την κυρία Γκούτελαντ, το ερώτημα της κυρίας Γκούτελαντ, θα πρέπει να σας δώσω την ίδια απάντηση σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Το θέμα είναι άκρος ενδιαφέρον, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και ε, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι θέμα δικής μας αρμοδιότητας. Περιμένουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα λάβουμε θέση και εμείς. Σε σχέση με την νόμιμη πρόσβαση στα φάρμακα, εδώ μιλάμε ιδιαίτερα για τα φάρμακα αντιμετώπισης των νεοπλασιών. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας, η πρόσβαση δηλαδή, η ίση πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στις 14 και 15 Απριλίου. Αλλά πάντα μιλάμε για την ίση πρόσβαση στα φάρμακα. Αυτή είναι η εποδός μας. Um, Προς τον κύριο Πανασέσκου, νομίζω στο πρώτο σας ερώτημα απάντησα για το, ως προς το εργαστήριο της στην Κλούσνα Πόκα για τον εμβολιασμό. Θα δούμε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας και να σας υποσχεθώ ότι παραμένουμε ανοιχτοί σε υποδείξεις. Όλες οι υποδείξεις είναι ευπρόσδεκτες καθ' όλη τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας. Και μετά από το εξάμεινο αυτό να είσαστε υπερήφανοι και εσείς για το έργο της Ρουμανίας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και ελπίζω να ε, μας πλαισιώσετε σε αυτές μας τις προσπάθειες και να μας επισκεφτείτε. Σας ε, ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Υπουργέ, ε, και θα σας υποστηρίξουμε και πιστεύουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και μεταγενέστερα, μετατρέποντας το λόγο σε πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την έλευσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Uh, Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Έχουμε ε, καλέσει ε, την αρμόδια διευθύντρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είναι η κυρία Ολίκη και, ο κύριος Δακούντο από την ε, αρμόδια ε, Γενική Διεύθυνση DG Growth. Και χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία και την ε, κυρία Διευθύντρια, για να αρχίσουμε τη συζήτησή μας για το θέμα αυτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Αυτή τη φορά έφερα μια μικρή παρουσίαση PowerPoint για να μιλήσουμε για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ένα συνολικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις, ε, ε τους ενδυνοκρινικούς διαταράκτες, λέει η κυρία Γιούλιχερ. Ε, είναι γνωστή και ως στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ε, δεν θα μπω τώρα σε μεγάλες λεπτομέρειες τα επιστημονικά δεδομένα και στον ορισμό των ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ε, ένας ε, ορισμός του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και το πρόγραμμα για την αντίστοιχη ασφάλεια των χημικών ουσιών. Είναι τρία τα χαρακτηριστικά τους και σορευτικά ε, ανεπιθύμητες δράσεις, ε, επιρροή στις ορμόνες και σχέση αιτίου αιτιατού μεταξύ των δύο. Δηλαδή διαταράσσεται η ορμονική ε, λειτουργία, η λειτουργία του ορμονικού συστήματος και μάλιστα υπάρχει συσχέτιση των δύο. Αυτά θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσουν και να κοιτάξουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και σε περίπτωση που χρειάζεται αφού τα ταυτοποιήσουμε να τα ρυθμίσουμε κιόλας ποιο είναι το πλαίσιο και το ιστορικό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Αυτό ανάγεται στην αρχή της δεκαετίας του 90, ε, όπου άρχισαν να εμφανίζονται ανησυχίε σχετικά με τις ουσίες αυτές και ήδη από το 1999 ε, είχαμε μια κοινοτική στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που εφαρμόστηκε το τελευταίο διάστημα, τελευταία 20 ετία πλέον. Ε, ιδιαίτερα το 2013 με 2016 το θέμα αυτό ε, συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά εξέχοντα τρόπο με δύο ψηφίσματα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες αλλά και στο Συμβούλιο κατά αντιστοιχεία και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ε, τη χρηστή διαχείριση χημικών για την προστασία και του περιβάλλοντος εκτός από την ε, ανθρώπινη υγεία, δημόσια υγεία. Έκτοτε το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ υψηλά στις προτεραιότητες όλων και όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε το 2017 Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε κριτήρια για να ταυτοποιεί τους ενδοκρινικούς διαταράκτες υπό τη νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα και τα βιοκτώνα όπου έχουμε σαφή νομική εντολή και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να ε, εγκρίνει μια ανανεωμένη ή μια νέα στρατηγική. Η ανακοίνωση λοιπόν, ε, η οποία εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2018, ε, αφορά και ακολουθεί αυτή την προηγούμενη δέσμευση και αφορά τρεις τομείς κυρίως. Πρώτον, την επιστήμη των ενδοκρινικών διαταρακτών. Ιδιαίτερα κάνουμε μια απογραφή που βρισκόμαστε και ποιες δυνατότητες έχουμε να ελέγχουμε ποιες ουσίες και ε, πώς οι επιστήμονες ενημερώνουν εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις ε, το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πολιτική και την νομοθετική ρύθμιση μέχρι τώρα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ας πούμε ποια είναι η έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι δοκιμές γίνονται, ε, τι κατευθυντήριες γραμμές γίνονται, πώς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αντιμετωπίζει τους διαταράκτες αυτούς. Επίσης τι έχει γίνει στο επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας. Και το τρίτο σημείο, ίσως και το πιο ενδιαφέρον αλλά και στραμμένο προς το μέλλον, πώς προτίθεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ευρωπαϊκή πολιτική για τους διαταράκτες αυτούς. Ε, θέλουμε να βρούμε μια προσέγγιση συνεκτική και συνεπή σε όλες τις χώρες και σε όλα τα επίπεδα και μια προσέγγιση που να βασίζεται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, τα πιο ενήμερα και χωρίς αποκλεισμούς με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Πολύ σύντομα ε, θέλω να σας αναφέρω κάποια από τα βασικά σημεία ε, της ανακοίνωσης για την επιστήμη αυτή. Όπως σας είπα, η όλη συζήτηση ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 και περί τα τέλη της δεκαετίας εκείνης αυξήθηκαν τα στοιχεία που συνέδεαν ε, τις ουσίες αυτές με την ανθρώπινη υγεία, την πρόκληση νόσων ή την αρνητική επίπτωση που έχουν στην άγρια πανίδα. Άρα, τώρα με επιστημονικούς όρους ε, υπάρχει συμφωνία για πολλά θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει ορισμένα από αυτά, ιδιαίτερα το 2016 και 2017 επανειλημμένα εδώ και στην Επιτροπή σας. Για παράδειγμα, ορισμοί ε, ορισμός των ίδιων των ενδοκρινικών διαταρακτών. Υπάρχει ευρεία έτσι, συνένεση θα έλεγα γι' αυτό. Η ιδιαίτερη ευαισθησία που μπορεί να έχουν τα έμβρια ή έφηβοι, αυτό πια ε, είναι αναγνωρισμένο κοινό και κατανοητό. Επίσης υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους δρούν και επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα οι ουσίες αυτές, καθώς επίσης και το ζήτημα της έκθεσης σε μείγμα ενδοκρινικών ε, διαταρακτών, ότι μπορούμε να έχουμε μια λεγόμενη επίπτωση κοκτέιλ, δηλαδή συνδυασμό επίδρασης. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες αβεβαιότητες ως προς τη γνώση μας, ας πούμε, πώς ε, συμβάλλει η έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες ε, στην ανάπτυξη μιας νόσου. Δηλαδή, μπορεί να ορίσει κανείς ένα ασφαλές ανώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό ε, είναι θέμα συζήτησης αρκετά επίμαχο. Επίσης γνωρίζετε ότι ε, κυρίως υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών και την εποπτεία του ΟΣΑ, η κατόπιν πρωτοβουλία του ΟΣΑ, έχουν γίνει πολλές δοκιμές, έχουν αναπτυχθεί δοκιμές ε, για να ανοιχνεύουν ε, την παρουσία ενδοκρινικών διαταρακτών στον οργανισμό. Βέβαια δεν είναι πλήρη ακόμα αυτά τα συστήματα και οι μηχανισμοί. Έρχομαι τώρα στην ευρωπαϊκή πολιτική και στην νομοθεσία ε, και στα θέματα της έρευνας μέχρι τώρα. Ε, ε, από το 1999 πάνω από 50 έργα έχουν χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί καλύτερα για τις ουσίες αυτές από το, τα αντίστοιχα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ περίπου και στο πρόγραμμα Horizon 2020 ε, ε, δόθηκαν ε, επιπλέον 52 εκατομμύρια ευρώ και είχε προβλεφθεί επίσης χρηματοδότηση και από άλλα προγράμματα για να αναπτυχθούν μεθοδοί ανείχνευσης και δοκιμών. Και ιδιαίτερα κάποια έργα του ορίζοντα 2020 τις τελευταίες μέρες έχουν προχωρήσει αφού έχουν εγκριθεί και οριστεί. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση της έρευνας όλα αυτά τα χρόνια, αρκετά σημαντική. Και έρχομαι τώρα στο νομοθετικό σκέλος. Και εκεί είχαμε προοδευτική ε, ενημέρωση και επικαιροποίηση τις τελευταίες δεκαετίες του κεκτημένου μας σχετικά με τα χημικά ε, σκευάσματα, τις χημικές ουσίες και το σημερινό πλαίσιο το νομοθετικό αναγνωρίζεται παγκοσμίω ως από τα πλέον προστατευτικά. Ε, ε, και πάλι το έχουμε πει αυτό και το έχουμε δει ε, σε πολλούς τομείς ε, νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται παγκοσμίω. Η δική μας προσέγγιση βασίζεται σε υψηλού επίπεδου επιστημονική πραγματογνωμοσύνη ε, στη βαρύς αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κρατών μελών και επίσης λαμβάνουμε υπόψη την αρχή της προφύλαξης. Και ένα τελευταίο χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό ε, παρακολουθούμε και πώς εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη αυτή την νομοθεσία. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα, περιορισμούς, απαγορεύσεις με διάφορα νομικά πλαίσια και νομοθετικά υπάρχουν και ειδικέ διατάξεις ε, για τις ουσίες αυτές, τη νομοθεσία περί ε, φυτοφαρμάκων και βιοκτώνων, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα ύδατα, το ρίτς και τις ε, ιατροτεχνικές συσκευές. Επίση υπάρχουν και γενικές απαιτήσει που μας επιτρέπουν να δράσουμε, όπως έγινε ε, στην ε, νομοθεσία για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, για τα καλλιντικά κτλ. Ε, αναπερίπτωση, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει νομοθετική ε, δράση. Παραμένω στην νομοθεσία E Τι συμβαίνει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σε διάφορα επίπεδα για διάφορες δράσεις με στόχο να αναπτύξει μια οριζόντια προσέγγιση έτσι ώστε να ταυτοποιούνται οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Γιατί αυτή είναι η πρώτη πρόκληση, το πρώτο πρόβλημα, η ανέγνευση καν της ουσίας. Και μετά έχουμε στόχο να υπάρξει μια οριζόντια προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί ε, για τα φυτοφάρμακα και τα ε, βιοκτώνα το 2017. Επίσης, ε, ανανεώνουμε και κυριοποιούμε τα στοιχεία για να μπορούμε καλύτερα να ανοιχνεύουμε τις ουσίες αυτές και εκτιμούμε και αξιολογούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και την επικοινωνία στην αλυσίδα παραγωγής και στα ενημερωτικά δελτία να γνωρίζουμε ότι κάποιες ουσίες ε, υπάρχουν σε κάποια προϊόντα και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές οι ουσίες. Επίσης, έχουμε και επιπλέον μέτρα και εργαλεία και μέσα, κάποια είναι πιο οριζόντια, όπως είναι η πρόταση τωρινή για η νομοθεσία γενικά για τα τρόφιμα, για τη διαφάνεια και την βιωσιμότητα της ε, εκτίμησης του κινδύνου, συνομοθεσία για τα τρόφιμα. Άλλο παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά, ε, για τις συσκευασίες ε, ή η ενημέρωση του νομικού πλαισίου για την επαγγελματική υγιεινή ε, και ασφάλεια στην εργασία. Πώς έχει τώρα η διεθνή συνεργασία για να τελειώσω. Είναι και πολυμερή. Σας ε, μίλησα προηγουμένως για τον ΩΣΑ που είναι πραγματικά ένα σημαντικό βήμα για να έχουμε ανάπτυξη διεθνώς συμφωνημένων δοκιμών αλλά υπάρχουν και άλλα πολυμερή φόρα όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το πρόγραμμα του περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Διμερή συνεργασία τώρα έχουμε ε, για το θέμα αυτό ε, με κάποιες χώρες όπως είναι τρίτες χώρες φυσικά, οι Ηνωμένε Πολιτείε. που το βλέπουν με το ίδιο μάτι. Εμάς οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Κίνα για να σας αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα κρατών. Τώρα, για το κομμάτι της ανακοίνωσης που κοιτάει προς το μέλλον τώρα. Για τη μελλοντική πολιτική της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν εξακολουθεί να είναι προσιλωμένη στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Και επιθυμεί να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά σίγουρα χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα. Μέσω της στρατηγικής αυτής προσέγγισης θέλουμε να βασιστούμε στην εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης πάντοτε χαρακτηρίζει τις αποφάσεις μας. Στόχος μας είναι να τα εξή, οι εξή στόχοι, να ελαχιστοποιήσουμε την συνολική έκθεση στους ενδοκρινικούς διατράκτες, να επιταχύνουμε την ανάπτυξη μιας ερνητικής βάσης, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουμε στη γνώση και να προωθήσουμε τον ε, διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ μας δράσεις, έχουμε αναλάβει να ε, κάνουμε ένα fitness check, οριζόντιο fitness check για τους ενδοκρινικούς διαταράκτε. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικές ε, ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωση. Έχουμε απουσία οριζόντιων κριτηρίων για παράδειγμα, έχουμε διαφορετικές νομοθετικέ ρυθμίσεις για τους διαφορετικούς νομοθετικούς διαταρακτέ. Είναι για πρώτη φορά που θα εξετάσουμε λεπτομερώς, θα βάλουμε κάτω από το μεγεθυντικό φακό την νομοθεσία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάρουμε επίσης πληροφορίες από μελέτες και θα χρησιμοποιήσουμε και δεδομένα που ήδη έχουμε από την αξιολόγηση που έχει ήδη γίνει, που λαμβάνει η χώρα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση της οδηγίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ε, θα ξεκινήσουμε ε, με ένα οδικό χάρτη που θα μπει σε διαβούλευση για τρεις μήνες. Ε, θα έρθουμε σε επαφή και διαβούλευση με τους όλους ενδιαφερόμενους και όλα αυτά θα ξεκινήσουν μέσα σε, στις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεύτερον, όπως είπα, θα αναζητήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχουμε. Ε, έχουμε αναλάβει την ευθύνη να κλείσουμε τα γνωσιακά κενά που έχουμε, το είπα αυτό και προηγουμένως, ακολουθώντας συγκεκριμένες ερευνητικέ κατευθύνσεις και με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Τρίτος στόχος, μια προσέγγιση που δεν θα αποκλεί κανέναν ενδιαφερόμενο. Θα συζητήσουμε με τους επιστήμονες, με το ενδιαφέρομενο κοινό, με τους εμπλεκόμενους γενικότερα. Θα οργανώσουμε ένα ετήσιο φόρουμ για τους διαγνωκλινιακούς διαταράκτες. Ε, η πρώτη συναντίαση του θα γίνει το μέσα στο 2019. Θα αυξήσουμε την στήριξή μας ε, στον ΩΣΑ, προκειμένου να ε, προωθηθεί η έρευνα στου διεθνούς, η δουλειά των διεθνών οργανισμών. Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε τη δυνατότητα οι ενδοκρινικοί διασταράκτε να συμπεριληφθούν στο υπάρχον διεθνέ σύστημα ταξινόμησης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούμε για άλλες κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Προετοιμάζουμε μια, ε, ένα, μια ε, σελίδα στο ίντερνετ θα είναι ενιαία θηρίδα για όλους τους ενδιαφέρονους και τους πολίτες που έχουν ανησυχίες για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και καθώς επίσης ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ειδικές, να εφαρμόσουν ειδικές πληροφοριακές και εκπαιδευτικές εκστρατείες. Η στρατηγική, όπως σας είπα, υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του περασμένου έτους, του 2018, και σύντομα θα ξεκινήσει η εργασία, ε, η εφαρμοστική διεργασία τις επόμενες ομάδες πιο συγκεκριμένα. Αυτά, εγώ και οι συναλφοί μου είμαστε έτοιμοι, οι συναλφοί μπορούν να σας μιλήσουν για τα, για τα καλλιντικά αν χρειάζεται. Ο κ. Δακούντο να μιλήσει πράγματι για τα καλλιντικά. θα συμπληρώσω τα όσα είπε η συνάδελφός μου. Ο κανονισμός για τα καλλιντικά απαιτεί να ε, ξαναδούμε τα προϊόντα τα οποία έχουν ε, ιδιότητες ενδοκρινικών διατρακτών και περιλαμβάνονται στα καλλιντικά ε, υιοθετήθηκε αυτή η, αναθεω, η έκθεση την ίδια μέρα που υιοθετήθηκε και το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε η συναλφός μου προηγουμένως. Ο κανονισμός δεν έχει ε, ειδικέ διατάξεις για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Υπάρχει όμως ένα σύνολο μέτρων, εφαρμοστικών μέτρων, τα οποία υιοθετήθηκαν για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης ενδοκρινικών διαταρακτών στον τομέα των καλλιντικών. Με στόχο την υψηλή επίπεδο προστασία της ανθρωπινής υγείας. Αυτές οι ουσίες ε, περιορίζονται ή απαγορεύονται είτε επειδή είναι τοξικές ε, καρκινογενείς ή μεταλλαξιογόνες ή σε άλλες περιπτώσεις επειδή υπόκειται σε ιδιαίτερα μέτρα, ειδικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση ε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μετά από μια αξιολόγηση κινδύνου που κάνει Ευρωπαϊκή πολιτική, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Πολιτών για την υγεία των πολιτών ε, και μετά από μια ειδική μελέτη για τους ενδοκρινικούς διαταρακτούς του 2014 ε, λαμβάνοντας υπόψη και τον ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση που γίνεται συστηματικά από την Επιστημονική Επιτροπή, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες θεωρούνται ως ουσίες που δημιουργούν ανησυχίες για την ανθρώπινη υγεία και εξετάζεται η έκθεση συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όπως παιδιά ή έγκες γυναίκες σε αυτές τις ουσίες. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης. Δύο κυρίως. Πρώτον, ότι ο κανονισμός καλλιντικών μέχρι τώρα ήταν το κατάλληλο εργαλείο για την διαχείριση αυτών των ουσιών που μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οπότε έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να παίρνουμε, να λαμβάνουμε τα κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, βασιζόμενοι στα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε. Δεύτερο συμπέρασμα, ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον με απαγορεύσεις ανδροκρινικών διαδρακτών στα καλλαντικά. Ήδη έχουν, ήδη η έκθεση ανακοινώνει τέσσερα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι ότι η Κομισιόν θα καταρτήσει ένα κατάλογο ε, ενδοκρινικών διαταρακτών που ενδεχομένως αποτελούν κίνδυνο και δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από παγορεύσεις που προκύπτουν με βάση τον κανονισμό καλλιντικών. Αυτό ε, ξεκινάει με μια πρώτη λίστα ουσιών στην ομάδα εργασίας των καλλιντικών, κάτι που μια, ένας κατάλογος παρουσιάστηκε ήδη στο Δεκέμβριο του περασμένου χρόνου στα κράτη-μελικές τους ενδιαφερόμενους η Επιστημονική Επιτροπή θα εμπλακεί στη συζήτηση αυτού του καταλόγου. Το δεύτερο βήμα είναι όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κατάλογος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 η Κομισιόν θα, ε, ξεκι, θα ζητήσει ε, από τους εμπλεκόμενους και από τον ακαδημαϊκό κόσμο ε, περισσότερα στοιχεία για αυτές τις ουσίες, δεδομένα. Ε, από τα δεδομένα τα οποία θα συλλεγούν, θα, η Κομισιόν θα προετοιμάσει εντολές στην Επιστημονική Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση ασφάλειας αυτών των ουσιών και τέταρτο βήμα θα είναι το προφανές υπό το φως των αξιολογήσεων αυτών, στις οποίες θα προβεί η Επιστημονική Επιτροπή, η Κομισιόν θα υιοθετήσει όπου θεωρηθεί απαραίτητο όλα τα μέτρα που θα χρειάζονται. Δηλαδή εφαρμοστικές ε, κανονιστικές πράξεις για τον περιορισμό της χρήσης ή την απαγόρευση αυτών των ουσιών. Ευχαριστώ. Λέει πρόεδρος. Συνάδελφοι, σε εσά ο λόγος. Κύριος Μπότς. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε λέει ο ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό ε, των ενδοκρινικών διαταραχών και θέλει να βελτιώσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε σήμερα και να ρυθμίσει εγκάρσια στην νομοθεσία μας ε, τις ουσίες αυτές για να μπορούμε είτε να τις απαγορεύουμε είτε να περιορίζουμε τη χρήση τους. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, κατά την άποψή μου, δεν είναι η στρατηγική για την οποία έχει απευθύνει η έκκληση εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στρατηγική σημαίνει κάτι άλλο. Εγώ θα περίμενα περισσότερα πράγματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, πιο χειροπιαστά στοιχεία ε, συγκεκριμένα στοχευμένα κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Μητροπή φαίνεται να μην θέλει να αλλάξει τη σημερινή πρακτική ε, όπου ο ανθρώπινος οργανισμός ε, εκτίθεται για μακρύ χρονικό διάστημα σε μικρές ποσότητες επιβλαβών ουσιών. Αυτά όμως δεν συνάδουν με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα που έχουν αποδείξει ότι ακόμα και μικρές ποσότητες μπορεί να είναι πάρα πολύ ε, και μικρή συγκέντρωση, δηλαδή πάρα πολύ επιβλαβή, ιδιαίτερα σε ευάλωτε ομάδε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θέλει να διοργανώσει μία πάγια διάσκεψη, τακτική δηλαδή, ε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για περισσότερες συνέργειες κτλ. Ωραία όλα αυτά, αλλά κάτι δεν καταλαβαίνω και θέλω να μου εξηγήσετε. Τι περιμένετε να βγει δηλαδή από αυτό το φόρουμ. Πώς θα οργανωθεί ο διάλογος, ποιοι θα συμμετέχουν εκεί. Μη κυβερνητικέ οργανώσει, μη κερδοσκοπικέ οργανώσει, ο κλάδο, η βιομηχανία και με ποια θέματα θα ασχολούνται. Διότι έχω τον εξή φόβο μήπως είναι ένα απλό βήμα συζητήσεων όπου θα συζητούν οι πυρογνώμονες και οι ενδιαφερόμενοι και θα συζητούν και θα συζητούν χωρίς να βγαίνει τίποτα, κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, χωρίς να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να μου πείτε πολύ συγκεκριμένα αυτό το φόρουμ πώς θα λειτουργεί και τι θα κάνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ παρόντες. Ε, ε, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για ε, ενδεχόμενες θανατηφόρες αρρώστιες από τις ουσίες αυτές και υπάρχουν παντού ε, παιχνίδια στα ρούχα, σε μπουκάλια, σε πλαστικά ε, συσκευασίες ε, τροφίμων και δεν μας προστατεύουν οι διεθνείς νομοθεσίες. Ε, περιμένουμε εδώ και χρόνια ε, συγκεκριμένα κριτήρια και στρατηγική για όλες τις ουσίες αυτές και δυστυχώς σήμερα εγώ δεν άκουσα κάτι που να μου διασκεδάσει αυτές τις ανησυχίες. Έρχεται και μας τάζει ένα φόρουμ τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πού είναι η φιλόδοξη στρατηγική, που, πουθενά. Ανακοίνωση λέει, διάλογο, ε, καθοδήγηση και κατάρτιση για τους διαχειριστές κινδύνου αυτό που τους νοιάζει πιο πολύ είναι εσωτερική αγορά και λιγότερο υγεία ανθρώπων και ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα στις ε, έρευνες, στην επιστημονική έρευνα και τις μεθόδους δοκιμών εγώ ρωτάω πώς θα ταυτοποιούνται αυτές οι ουσίες και πώς θα απομακρύνονται από την αγορά. Συγκεκριμένα στα φυτοφάρμακα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εκεί άρχισε τα βιοκτώνα και τα φυτοφάρμακα. Το 2015 ήδη υπήρξε νομοθεσία ε, ε, για να ε, απαγορεύονται κάποιες ουσίες, αυτές οι καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή και μεταλλαξιογόνες αλλά ε, παρόλα αυτά ε, διαδικαστικά παρατείνεται η κυκλοφορία για τη μοξιστροπίν, χλώρο το νερό και τρία κλοπίτ που ξέρουμε ότι είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες. Ε, κυκλοφορούν ακόμα στην αγορά παρόλο που εδώ και καιρό έχει αποδειχθεί πόσο επιβλαβής είναι. Πότε θα μας προστατεύσετε επιτέλους από τις ουσίες αυτές και πότε θα τις αποσύρετε από την αγορά. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Γκούτελαντ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευκαιρία που μας δίνει να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα. Τίνω να συμφωνήσω με τις ανησυχίες των συναδέλφων. Αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν είναι αρκετά ή δεν είναι αρκετά στεναρά έχουν αποδείξει οι επιστήμονες σε διάφορες εκθέσεις και επιστημονικά πεδία, έχουν αποδείξει, λέω, ότι ενδοκρινικές, ε, ε, αυτές οι ενδοκρινικοί διαταράκτες επηρεάζουν τις ευάλωτες ομάδες. Για παράδειγμα, τις εγγύους, όπου το έμβριο εκτίθεται πάρα πολύ σε αυτό το κίνδυνο. Και δεν βλέπουμε α, αντίδραση. Ενώ υπάρχει συσχέτιση ε, των ουσιών αυτών με ασθένειες. Και επίσης πολλές ε, ε, από τις ε, νόσους που βλέπουμε σήμερα, καρκίνη, καρκίνοι, διαβήτης, συνδέονται με αυτά τα πράγματα, ακόμα και η ίδια και η ανάπτυξη του εγκεφάλου η κεφαλική ε, ανάπτυξη. Επίσης, τώρα τι μας λέτε, ότι θα κάνουμε συζητήσεις, θα πάρουμε κάποια μέτρα. Ε, τι κάνουμε, απλώς παρατείνουμε τη διαδικασία και τη διονίζουμε. Θα πρέπει η αρχή της ε, προφύλαξης να εφαρμόζεται με χειροπιαστά απτά αποτελέσματα. Πότε θα φέρει πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφές χρονοδιάγραμμα και μέτρα, όπως είναι αυτά που λέει η έκθεση. Και στη συνέχεια, γιατί η έκθεση δεν κάνει λόγο για τη μελέτη αντικτύπου. Τα καλλιντικά υποτίθεται είναι τομέας προτεραιότητας. Και ένα τελευταίο, αλλά σημαντικό, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου νομοθετικές αλλαγές για τα καλλιντικά, παρά το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρει κάποια στοιχεία. Και θα πρέπει να έχουμε διατάξεις παντού στην νομοθεσία για τις ενδο, τους διαταράκτες, ιδιαίτερα στα καλλιντικά. Αυτό γιατί δεν υπάρχει. Θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα να επιταχύνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη δημόσια υγεία. Κύριο Σεκχαουτ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και <laughs> την Επιτροπή για την παρουσίαση. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση σας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίπονο θέμα που σας αποσχόλησε εδώ και δύο χρόνια. Είπατε, μιλήσατε στην παρουσίαση για τα δύο κριτήρια. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσουμε την επταετία με δικαστικές υποθέσεις, δικόγραφα κλπ. Φυσικά κανένας δεν μπορεί να το ξεχάσει και ελπίζω μην το έχει ξεχάσει και η Κομισιόν για να ε, φτάσει σε κάτι πιο απτό, διότι υπάρχουν ε, πολλά βιομηχανικά συμφέροντα, γι' αυτό και άργησε χαρακτηριστικά η Επιτροπή. Όταν τον Νοέμβριο λοιπόν φτάσατε σε μία στρατηγική, ε, ίσως ε, φανταστήκατε ότι θα θεωρήσουμε ότι η Επιτροπή το παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα. Όταν δούμε αυτή τη στρατηγική, ο Θεός να την κάνει, βλέπω ότι μιλάμε για fitness ε, checks, φόρα διάφορα, ε, μια επικοινωνιακή τακτική και λοιπά. Αυτό που προτείνατε στο 7ο περιβαλλοντικό ε, πρόγραμμα θα έπρεπε να αποτελεί μια νομοθετική πράξη. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και ήθελα να μας πει η Επίτροπη πότε θα αποφανθεί για θέματα που είχε ε, υποσχεθεί ως συνομοθέτη στο 7ο πρόγραμμα, περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να φτάσει σε ένα μη τοξικό περιβάλλον μέχρι το 18, δηλαδή πέρσι. Άρα αθετήσαμε αυτό το ορόσημο, καθώς και ελαχίστο ποιήση έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μα πότε θα γίνει αυτό. Θα ακολουθήσει το νόμο επιτέλους η Επιτροπή. Μέχρι το 20 όλες οι ουσίες και αυτές που έχουν ε, στοιχεία που στοιχεία ενδοκρινικών διαταρακτών βρίσκονται στον κατάλογο REACH, αλλά θα έπρεπε να απαλληφθούν πολλοί από αυτούς. Τι θα κάνει η Επίτροπη μέχρι το 2020. Μέχρι το 20 επίσης θα πρέπει σε όλα τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθούν ε, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ε, τώρα όμως φτάσατε σε ε, απαγορεύσεις για φυτοφάρμακα και βιοκτώνα. Δηλαδή αυτό το κάνατε οριζόντια και μιλάτε για fitness checks και στα καλλιντικά φαίνεται ότι λέτε ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, δηλαδή υπηρετεί τις αξίες που προβάλλεται αλλά είχατε πει ότι μέχρι το 20 θα γίνει ένας άλλος ειδικό έλεγχος για τα καλλιντικά. Τώρα δηλαδή θα κάνετε ένα διαφορετικό έλεγχο καταλληλότητας για τα καλλιντικά. Δεν το παίρνετε λοιπόν στα σοβαρά και όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι το 20. Γιατί δεν έγιναν αυτοί οι έλεγχοι καταλληλότητας χρόνια πριν και γιατί τι είναι ε, στην ουσία ένα πρόκριμα για καθυστέρηση με βάση το 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αποφάσισαν οι αποκοινού νομοθέτες. Ε, η Κομισιόν θα πρέπει να φτάσει σε αξιόπιστες απαντήσεις και όχι να οργανώνει άλλο ένα φόρουμ όπου θα μιλήσουμε με τους εμπλεκόμενους φορείς και ούτω καθεξής. Ωραία, σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν και το πρώτο μέρος της συζήτησης. Τώρα, τι έχει να μας πει η Κομισιόν. Ποιος θα λάβει το λόγο. κυρία Λίκαρ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο ξανά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω στις πολύ συγκεκριμένες. Καταρχήν για το ετήσιο φόρουμ το μοντέλο μας δεν θα έχει αποκλισμούς, θα, είναι, θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων. Ένα φόρουμ στο οποίο θα μπορούν να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές, θα μπορεί να μάθει ο ένας από τον άλλο. Οπότε, ναι, πρόκειται για φόρουμ προβληματισμού, συζήτησης, το έχουμε δει όμως και αλλού, τέτοιου είδους ε, φόρουμ ε, δίνουν το ρυθμό και την, το έναυσμα για δράση, ε, νομοθετική δράση. Τώρα, πρόκειται για, για μια ανακοίνωση και ας ξεκαθαρίσω ότι σε όλη τη δουλειά που κάνουμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες έχει καταστεί σαφές ότι ορισμένες δυσκολίες σχετίζονται με ελλείψεις που έχουμε στο επιστημονικό μέτωπο. Με άλλα λόγια, δεν καταλαβαίνουμε όλα τα φαινόμενα. Και πολλά από τα σχόλια που έγιναν πριν από λίγο σχετίζονται με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, εξηγήσει κλπ. για τα ίδια θέματα. Για το ποια είναι η επίδραση των ενδοκρινικών διαταρακτών πιο συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες ασθένειες όπως ο διαβήτης κλπ. Μακάρι, θα έλεγα εγώ, να είχαμε προχωρήσει πιο πολύ επιστημονικά. στόχος είναι να πάρουμε αποφάσεις και κανονιστικές αλλά και μελλοντικά νομοθετικές. Έτσι ώστε και μάλιστα αυτές οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια. Δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Γι' αυτό το λόγο ε, κατευθύνουμε χρηματοδότηση στην έρευνα για να καταλάβουμε καλύτερα τη σχέση αιτίου αιτιατού και εδώ αλλά και αλλού σε άλλα σημεία της διαδικασίας. Τώρα, γιατί δεν έγινε μελέτη αξιολόγησης, μελέτη αντικτύπου, συγγνώμη. Να σας το εξηγήσω. Ο έλεγχος νομοθεσίας αυτό το fitness check, είναι ένα πρώτο βήμα. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε κάτι τέτοιο οριζοντίως σε όλους τους τομείς πολιτικής. Και θα προχωρήσουμε γρήγορα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θέλουμε να έχουμε πλέον μια σαφή εικόνα για το τι κάνει το ισχυρό ε, κανονιστικό πλαίσιο. Αν πετυχαίνει τους στόχους του, αν όχι, ή αν θα τα καταφέρουμε μόνο αν το τροποποιήσουμε. Και εκεί θα κάνουμε και τη μελέτη επιπτώσεων. Οπότε, γιατί ξεκινήσαμε από τα βιοκτώνα και τα παρασιτοκτώνα, γιατί αυτή ήταν νομική μας υποχρέωση καταρχήν. Αλλά ακόμα και σε δύο τομείς όπως αυτή που ήταν αρκετά σαφώς διαγεγραμμένη δυσκολευτήκαμε να καθορίσουμε κριτήρια τα οποία πραγματικά να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και να είναι βιώσιμα για το μέλλον. Οπότε το fitness check είναι το πρώτο βήμα και η επόμενη κομισιόν θα έχει χρόνο να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Αν αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω κανονιστικές δράσεις, νομίζω ότι τότε θα γίνει και η μελέτη αντικτύπου. Τώρα, αν έχουμε πάρει μέτρα για ουσίες που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, για τους τομείς που ξέρω εγώ περισσότερο, αλλά και πιο πέρα, στο ρίτσα ας πούμε, μπορώ να πω ναι, έχουμε πάρει μέτρα. Τα... Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε αποσύρει από την αγορά πολλά προϊόντα τα οποία είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες. στόχος της Κομισιόν και με τα καινούργια κριτήρια που υιοθετήσαμε για τα βιοκτώνα και τα παρεστοκτώνα ε, είναι αυτός ακριβώς. Αλλά βέβαια τα κριτήρια μας θα πρέπει με τη στήριξη της επιστήμης να γίνουν πιο ακριβή καταλαβαίνοντας καλύτερα την αιτία και το αποτέλεσμα. Έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα για περισσότερες ουσίες αν εντοπιστούν και κατονομαστούν ως ε, ενδοκρινικοί διαταράκτες. Για τα παραστοκτόνα και τα βιοκτόνα, όπως είπε και ο πίτροπος Αντροϊκάητης, ε, αρχίσαμε να εφαρμόζουμε αμέσως τα καινούργια κριτήρια και θα, πάρουμε, θα αναλάβουμε δράση αν εντοπιστούν ουσίες που έχουν τέτοιου είδους επίδραση στον οργανισμό. Η οριζόντια προσέγγιση σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε στο fitness check. Το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οριζόντια προσέγγιση δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνατότητα να αναλαμβάνουμε δράση. Νομίζω ότι πολλοί από εσά γνωρίζετε τι έχουμε κάνει για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες σε ένα αριθμό από ε, κανονιστικούς ε, ε, πυλώνες. Τώρα για τη δυσφενόλη α. Την δυσφενόλη α την περιορίσαμε στα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε μεγάλο βαθμό και μέσα στο 18 ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να εξακολουθήσει να εξετάζει την ουσία αυτή και εδώ πάλι χρειαζόμαστε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία αν, χρειάζεται, αν προκειμένου να ε, προχωρήσουμε σε πιο αυστηρά μέτρα. Σε οτιδήποτε έχει σχέση με την δημόσια ασφάλεια, ε, προφανώς ε, ε, η δημόσια ασφάλεια έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Ο συνάδελφός μου, θέλετε, δεν μπορούσε να απαντήσει για τα καλλιντικά, σε περίπτωση που το επιθυμείτε. Ναι, ευχαριστώ. Σύντομα σας παρακαλώ. Uh, uh, ναι, έγινε μια ερώτηση γιατί δεν προβλέπουμε ε, αλλαγές, τροποποίηση στον κανονισμό για τα καλλιντικά. Παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός αυτός δεν αναφέρεται ε, ρητά σε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να επιβάλλουμε απαγορεύσεις ή περιορισμούς στη χρήση των ουσιών αυτών. Δεν υπάρχει νομικό κενό. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κανονισμός. Έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας όλα τα εργαλεία για να πάρουμε ό,τι μέτρα χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε υψηλή προστασία. Βέβαια, τούτου λεχθέντος, ο κανονισμός και τα καλλιτικά θα ενταχθεί στην οριζόντια διαδικασία, την εγκάρσια στη νέα στρατηγική. Ευχαριστώ. Okay, this concludes this item and... Uh, Μάλιστα, τελειώνει αυτό το θέμα. Η κυρία Χάζεκαμπ ζητεί το λόγο. Κοιτάξτε, έχουμε καθυστέρηση, 15 λεπτά τουλάχιστον. Αυτά δεν ήταν απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει, λέει ο κύριο Εκχάουτ. Θα πρέπει να μα παίρνει σοβαρά υπόψη η Κομισιόν. Έκα... Μισό λεπτό, κύριε Εκχάουτ. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Να μα πείτε σε τι δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημόσια αλλά δεν θα ξαναδώσω το λόγο στην Επιτροπή που δεν απάντησε στις ερωτήσεις, γιατί έχουμε καθυστέρηση. Και η κυρία Χάζεκαμπ, παρακαλώ, κάτω από δύο λεπτά έκαστο. Ο κύριο Σέικχαουτ. μα δεν μα απάντησαν συγκεκριμένα για την στρατηγική τη Ένωση για ένα μη τοξικό περιβάλλον που υποτίθεται ότι θα είχαν φέρει μέχρι το 18. Ούτε κουβέντα δεν μα είπαν για ποιο λόγο, γιατί καθυστέρησε και πότε θα έρθει. Πώ θα εξασφαλίσουν ότι όλες οι ουσίες που μας ανησυχούν τόσο πολύ θα μπουν στο κατάλογο του REACH που υποτίθεται θα γίνει μέχρι το 2020 και σε όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι ουσίες ε, μέχρι το 2020 και όλες αυτές οι δράσεις για την ασφάλεια ή η, η, ε, θα καθυστερήσουν τόσο πολύ, θα ξαναχάσουμε και την προθεσμία του 2020, όπως έχουμε χάσει όλες τις προθεσμίες μέχρι σήμερα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και θέλω πραγματικά να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεσμεύονται να τηρήσουν αυτές τις προθεσμίες, διότι είναι και ευευλημένες δια νόμου. Μάλιστα. Σας ακούσαμε. Από την πρώτη φορά το είχατε ξεκαθαρίσει αυτό. Επέλεξαν να μην απαντήσουν. Η κυρία Γιούλη έχει απάντηση γι' αυτό. Λοιπόν, για τη στρατηγική που λέτε για το τοξικό περιβάλλον. Ε, προφανώς δεν έχει έρθει ακόμα, μπορώ να το επιβεβαίωσω. Ε, μας προβληματίζει και το συζητάμε στις υπηρεσίες μας, ιδιαίτερα για να προετοιμαστούμε για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι καθοδόν το θέμα, έχει δρομολογηθεί. Για το REACH δεν ξέρω, δεν δουλεύω εγώ για το REACH αλλά συνεχώς επεξεργάζονται τη λίστα υποψηφίων ουσιών προς προσθήκη. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι 180-90 ουσίες που ε, αναθεωρούνται στο REACH. Ε, μπορεί να μας βοηθήσει άλλος συνάδελφος, συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω αυτό, τουλάχιστον, όσο μπορώ. Έχω την τελευταία έκθεση ε, της ΕΧΑ, του οργανισμού, για τα χημικά ε, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2018 και αφορά το διάστημα μέχρι το 2020. Κάθε χρόνο ελέγχει αυτός ο οργανισμός τις χημικές ουσίες που έχει στην τράπεζα δεδομένων του, τις ε, ε, ουσίες που έχουν κατοχωριστεί και σε άλλες τράπεζες δεδομένων που έχουν καταγράψει ΜΚΟ, συνδικάτα και γίνεται ο έλεγχος. Γράφει στην έκθεση ο Οργανισμός για τα Χημικά ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2018 έχουν ανοιχνεύσει 1.699 ουσίες ως ενδεχομένως ανησυχητικές. Δεν είναι όλες αυτές οι ουσίες ενδοκρινικοί διαταράκτες. 377 περίπου και ο Οργανισμός για τα Χημικά τις μελετάει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι περισσότερες από τις ουσίες αυτές τον Απρίλιο του 2018 δεν ήταν ενταγμένες στο REACH, δεν είχαν αυτή την καταχώρηση, περίπου το 60% των ουσιών. και από τις 377 που είναι ενδεχόμενοι ενδοκρινικοί διαταράκτες, το 1 τέταρτο έχει ρυθμιστεί, ενώ οι υπόλοιπε, ε, μάλλον άλλο ένα 10 με 15% μελετάται αυτό τον καιρό και ορισμένες από τις άλλες ύποπτες ε, απεδείχθη ότι δεν είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Από τις 377 λοιπόν δεν έχουμε καταλήξει στο να υπάρχουν κάποιες ουσίες που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και δεν ξέρονται. Και πέρσι το καλοκαίρι έβγαλε αυτή την ανακοίνωση η ΕΧΑ, ο Οργανισμός Φαρμα... Ε, Χημικών, συγγνώμη, που κάθε χρόνο κάνει μελέτες. Μάλιστα, εδώ ολοκληρώνεται το θέμα αυτό για σήμερα. Όχι, λέει η κυρία Χάζα, κάνω εγώ ζητώ το λόγο τόση ώρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ. Λυπάμαι πάρα πολύ σας είπα ότι έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, 20 λεπτά. Δεν γίνεται να σας ξαναδώσω το λόγο. I'm sorry, you... Ζητώ συγγνώμη, μου είπατε ε, να επαναλάβω την ερώτηση μου, που ήταν και μικρή. Γιατί δεν περίμενα και πάρα πολλά, ούτε ε, προσδοκούσα να μου δώσουν συγκεκριμένη απάντηση. Θέλω να την επαναλάβω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Χάζευ, παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτησή σας. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ. Θα τα πω Ολλανδικά. Άρα, εγώ περίμενα για να μου απαντήσετε για τις τρεις συγκεκριμένες ουσίες ε, το 2005 και 2006 κυκλοφόρησαν στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι δηλητήρια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και δεν θα έπρεπε να τους είχε δοθεί έγκριση. Παρ' όλα αυτά το 2016 δόθηκε παράταση για ένα χρόνο και το 2017 πάλι παράταση για ένα χρόνο και το 2018. Είναι τρεις ουσίες αυτές που τρία χρόνια κυκλοφορούν παρόλο που είναι αποδεδειγμένα ενδοκρινικοί διαταράκτες και θα έπρεπε να απαγορεύονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει και στο κανονισμό για την προστασία των φυτών ότι πρέπει να απαγορευθούν και στη νομοθεσία για τα τρόφιμα. Και σας ρώτησα πότε επιτέλους θα απαγορευθούν αυτές οι ουσίες στην Ευρώπη. Είναι σκέτο, σκάνδαλο και έσχος που ακόμα επιτρέπονται. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα για τρίτη φορά. Και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σφάρτς που είναι εισηγητή της ευρωπαϊκή Οικονομικής ε, και Κοινωνικής Επιτροπής για την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία, για την ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τα ύδατα και τα απόβλητα από την ΕΟΚΕ. διερευνητική γνωμοδότηση κατέρτισαν, εκπώνησαν για τη δική μας επιτροπή. Τους το είχαμε προτείνει εμείς και ε, ε, με χαρά τη δέχτηκα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σφάρτς που είναι εισηγητής και θέλουμε να ακούσουμε τα συμπεράσματά σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εξ ονόματος της ΕΟΚΕ σας εύχομαι καλή χρονιά για το 2019 και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την ανάθεση στην ΕΟΚΕ σε σχέση με τη διερευνητική γνωμοδότηση για την ε, ε, ποιότητα την περιβαλλοντική νομοθεσία στους τομείς της μειότητας του αέρα, των υδάτων και των αποβλήτων. Οι συζητήσεις μπορεί να είναι αρκετά ζωηρές, όπως είδαμε και με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, γιατί το διακύβευμα είναι η υγεία των πολιτών αλλά και των οικοσυστημάτων γενικότερα, χωρίς τα οποία καμία οικονομία δεν είναι βιώσιμη μακροχρόνια. Και αυτό ανακύπτει από τη γνωμοδότηση αυτή. Υπενθυμίζουμε ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης με, ε, μέσα στα πλαίσια του ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες είναι πολύ απαιτητικοί σε θέματα περιβάλλοντος και για να υπάρχει αξιοπιστία στα θεσμικά όργανα πρέπει να αποδίδουμε και να φτάνουμε σε ε, αποτελέσματα. Άρα είναι θέμα της δικής μας αξιοπιστίας να τηρήσουμε αυτό το νόμο, ο οποίος έχει εγκριθεί και ο οποίος ε, τελειοποιήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι θέμα αξιοπιστίας για να υπάρχει ίση ε, αντιμετώπιση και ικανοποιητική, έτσι ώστε οι πολίτες να εμπιστεύονται την Ευρώπη ως προς τα, περιβαλλοντικά, αλλά και επειδή σε οικονομικό επίπεδο έχει νόημα να τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία υπέρ του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά κέρδη οικονομικά στο τομέα του ανταγωνισμού και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος Βέλλα πρόσφατα είπε ότι μιλάμε για 500 ε, δις ετησίως, ε, τα οποία αποταμιεύουμε αν εφαρμόσουμε το περιβαλλοντικό δίκαιο. Αυτό είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το δίκαιο, αυτή τη νομοθεσία για να μην δημιουργούνται και αδικίες. Εκεί που υπάρχουν αδικίες και ανισότητες υπάρχει και απώλεια αξιοπιστίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έτσι έχει λοιπόν αυτή η διερευνητική γνωμοδότηση, ανέκυψε μετά από γνωμοδότηση, μετά από ανακοίνωση, την ανακοίνωση υπαριθμών 10 το 2018 της Επιτροπής που αφορά ένα πρόγραμμα δράσης για την νομοθεσία για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, από την οποία ε, ανασύραμε πολλά αποτελέσματα, συμπεράσματα και γι' αυτό φτάσαμε σε πολλά παρόμοια συμπεράσματα. Θα σας τα αναφέρω εντάχει για να υπάρχει χρόνος για ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Χαιρετήσαμε ως ΕΟΚΕ τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για και την ανακοίνωση σε σχέση με τη διακυβέρνηση του περιβάλλοντος καθώς και τη σχετική νομοθεσία. Όμως, όπως πολύ συχνά, προτείναμε ε, ορισμένες ιδέες για να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο. Πανηγυρίσαμε τα 50 μας χρόνια πέρσι ως ΕΟΚΕ και ξέρετε εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας των πολιτών, τους εργοδότες, τα συνδικάτα και τους πολίτες που συμμετέχουν σε διάφορες ενώσεις προστασίας ε, και του περιβάλλοντος, από οικογένειες, από διάφορους οργανισμούς και ενώσεις προστασίας και σε αυτή τη γνωμοδότηση φτάσαμε σχεδόν ομόφωνα. η οποία δείχνει έλλειψη βούλησης από κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία. Πολλές κυβερνήσεις λοιπόν δυστυχώς δεν μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το δίκαιο γιατί δεν υπάρχει σχετική θέληση. Ε, αυτό είναι πολύ σοβαρό αλλά έτσι έχει. Δεύτερον, υπάρχει έλλειψη πόρων κατά συνέπεια για να ε, τεθεί σε εφαρμογή το περιβαλλοντικό δίκαιο. Δεν υπάρχουν ε, χρηματικοί πόροι, ούτε και ανθρώπινοι. Θα πρέπει να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα τήρησης του νομοθετικού πλαισίου. Πώς ε, μπορεί να γίνει αυτό. Χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό για να κοινοποιήσει το περιβαλλοντικό δίκαιο, αλλά και για να ε, τεθεί σε εφαρμογή και να υπάρχει ένα κυρωτικό καθεστώς. Αυτά είναι και οι πρώτες μας ε, σκέψεις και συστάσεις και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μεταφέρουν αυτό το πλαίσιο στο πολιετές. Εκεί θα εγγραφούν οι πόροι για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών λόγω διαφορετικής αντιμετώπισης. Η ΕΟΚΕ μέσω των οργανώσεών της και των ευρωπαϊκών δικτύων κρίνει ότι μπορεί πράγματι να βοηθήσει με τα περιορισμένα της μέσα, αλλά οι οργανώσεις μας ε, έχουν έχουν επιτόπιους φορείς και πολίτες που επαγρυπνούν έτσι ώστε τα κράτη να ανταποκριθούν σε αυτό τους το καθήκον. Θα πρέπει να παρεμβαίνουν λοιπόν σε τακτά χρονικά διαστήματα και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει μία ε, γονομοδότηση η οποία μας ζητήθηκε μέσω του Αντιπροέδρου Τίμερμανς. Τώρα ως προς το θέμα του προσωπικού και των εγγεγραμμένων πόρων σχετίζεται με την τήρηση του περιβαλλοντικού δικαίου στους ε, συγκεκριμένους τομείς γενικότερα. Όχι μόνο εκεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά και γι' αυτό μιλήσαμε για αέρα, ύδατα και απόβλητα. Και ιδιαίτερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, επιθεωρητές περιβάλλοντος, όμως σε επίπεδο κρατών μελών θα είχε μεγάλη σημασία να γίνεται ειδική κατάρτιση μέσα στα πλαίσια και εισαγγελικών αρχών έτσι ώστε να μπορέσει να παρέμβει η δικαιοσύνη στα περιβαλλοντικά. Γιατί τι βλέπουμε το περιβαλλοντικό ως προς το περιβαλλοντικό δίκαιο. Εάν γίνει προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης των πολιτών, δυστυχώς το θέμα δεν γίνεται κατανοητό από τους δικαστές, διότι δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση. Άρα ε, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν καταλήλως. Δηλαδή, χανόμαστε σε διαφόρους ε, δεδάλους πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό χρειάζονται εξειδικευμένοι ε, εισαγγελείς. Θα ήθελα τέλος να υπενθυμίσω ότι χρειαζόμαστε τη σωστή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου έτσι ώστε να φτάσουμε και στους απότερους στόχους μας για τον ορίζοντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις συμφωνίες του Παρισιού. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτές τις ε, συμφωνίες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας αυτή. Ερωτήσεις? Καλώς. Κύριε Σουάρτς, να σας ρωτήσω εγώ. Το περιβάλλον είναι από τους τομείς εκείνους που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό προσφυγών επί παραλήψη στο δικαστήριο. Για ποιο λόγο, γιατί δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στους τομείς που καλύπτει η γνωμοδότησή σας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και θα μπορούσατε να μας πείτε και λίγα λόγια. Μήπως χρειαζόμαστε και δικαστές και εισαγγελείς που να ειδικεύονται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Να είστε δύο ερωτήσεις παρακαλώ αν θέλετε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτή με την οποία ξεκίνησα. Είναι ο πολιτιστικός παράγοντας αυτών που παίρνουν αποφάσεις. Οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων καταρχήν και αυτοί που τους φέρνουν στην εξουσία. γιατί πολύ συχνά δεν είναι οι ίδιοι οι πολίτες που τους ε, στέλνουν στην εξουσία. Είναι ένα ολόκληρο νομικό σύστημα που επιτρέπει την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και την διάδοση των ιδεών τους μέσω των μέσων ενημέρωσης. Αυτό αφορά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα μικρότερο βαθμό. Τα, οι περισσότερες αποφάσεις, τα, περισσότερα, τα μεγαλύτερα διακυβεύματα βρίσκονται στα κράτη-μέλη με επιχειρήσεις πίσω από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις με πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ε, και παρόλο ότι ε, δεν θα υφίσταται οικονομία σε ένα νεκρό πλανήτη, αυτό το αγνοούν, το αμελούν. Οπότε ο πολιτιστικός παράγοντας είναι ο πρώτος παράγοντας και αν δεν αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται οι θύνοντες θα τεθούν σε κίνδυνο οι ίδιες δημοκρατικές αξίες μας. Αυτό συζητείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, στο μέτρο που πλησιάζουμε και στις επόμενες ευρωεκλογέ. Οπότε το πιο μεγάλο, η πιο μεγάλη πρόκληση είναι η πολιτιστική. Χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για να υλοποιηθούν τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. αν αυτά τα δικαιώματα είχαν υλοποιηθεί, τότε πολύ λιγότεροι πολίτες θα κατέφευγαν στη δικαιοσύνη. Ας προσέχουμε λοιπόν ποιον ψηφίζουμε. Ε, ένας συνάδελφος το έθιξε αυτό. Ρώτησε την Κομισιόν επανειλημμένως, θα, θα ε, σεβαστείτε τους κανόνες που εσείς οι ίδιοι δημιουργείτε. Αυτά είναι θέματα ουσίας. Ας γίνουν πραγματικοί δημοκράτες που εφαρμόζουν τους νόμους που ψηφίζουν. Δεύτερευόντως, οι εξειδικευμένοι δικαστές και εισαγγελείς για θέματα περιβάλλοντος. Αυτές οι ιδέες δεν είναι μόνο δικές μας στην ΕΟΚΕ. Είναι και ιδέες του δικτύου Impel, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο από επαγγελματίες του κλάδου και που αντιλαμβάνονται ότι οι δικαστές δεν έχουν χρόνο να ειδικευθούν για τέτοιους, ε, σε τέτοιου θέματα και χρειάζεται διαρκώς να περνούν από ένα ζήτημα σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό. Χρειάζεται οι δικαστές να γνωρίζουν όχι μόνο την νομοθεσία, που τα νομοθετικά κείμενα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα σε αυτό το τομέα, αλλά πρέπει να γνωρίζουν και την προηγούμενη νομολογία και τις περισσότερες φορές τα άτομα αυτά δεν λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε στέρεα νομικά κριτήρια. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε εξειδίκευση. Ζητά το δίκτυο ΕΜΠΕΛ και εμείς γινόμαστε, ε, συμμεριζόμαστε μάλλον το αίτημά τους. Οι δικαστές χρειάζονται ειδίκευση, χρειάζονται χρόνο για να... και εμπειρία μεγάλη σε τέτοιου ζητήματα. Well, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σβάρτς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει τίποτα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Many thanks. Many thanks. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το αίτημα και υπήρξε και διερευνητική γνωμοδότηση. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με πολλά από τα ευρήματά της και ιδιαίτερα με τα γενικά σχόλια που αναφέρονται στο δεύτερο μέρος του κειμένου η ανάγκη να αποφύγουμε τις ε, αποκλίσεις και τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, τι δυνατότητες έχουν οι κυβερνητικοί μηχανισμοί, η ε, συνειδητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, σε όλα αυτά συμφωνούμε, είναι κρίσιμα και πολύ σημαντικά. Στόχος αυτής της ε, γνωμοδότησης δεν ήταν να επαναλάβει το γενικότερο έργο που είχε παραγάγει μέχρι τώρα η ΕΟΚΕ, δεν αναφέρονται κάποια στοιχεία που αναφέρονται στα γενικά κείμενα. Είναι πολύ σημαντικά για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, των υδάτων και των αποπλήτων. Προφανώς ε, δεν είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενθαρρύνουμε προς συμμόρφωση αρκετά. Χωράει η βελτίωση και στους τρεις τομείς. Πάντως υπάρχει βελτίωση και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι στα κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτά τα τρία, μερικές από τις συστάσεις έχουν να κάνουν μάλλον με αναθεώρηση των κειμένων ε, που ισχύουν των νομικών παρά ε, με την ε, εφαρμογή τους. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, βεβαίως. Μπορεί να χρειαστεί έλεγχος τη νομοθεσία για την καταλληλότητα, αλλά το θέμα είναι να εφαρμόζονται όπως έχουν. Υπάρχουν και δύο στοιχεία που θα θέλαμε να προσθέσουμε στην έκθεση αυτή. Το πρώτο είναι η σημασία της ε, ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης. Έχουμε δει ότι το σημαντικότερο τμήμα άλλων πολιτικών όπως είναι η ενέργεια, η γεωργία, ε, ε, οι μεταφορές, αυτή τα νετρικά, όλα αυτά είναι κάποιοι τομείς, άλλοι τομείς πολιτικής που έχουν όμως επίπτωση στο περιβάλλον. Και επίση η διαφάνεια και η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία. Πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό. Όταν δεν γνωρίζει ο κόσμος τι μπορεί να κάνει, τότε δεν μπορεί να δράσει και αποτελεσματικά. Ε, αυτή ήταν μια σύντομη απάντηση, έτσι, σύντομη εκδοχή της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σφάρτς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση αυτή και τα σχόλιά της. Ολοκληρώνεται εδώ το σημείο αυτό της ημέρης της διάταξης. On topic Τώρα τι θα γίνει με το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν βλέπω τον κύριο Ντόρτ. Λέγει ah, Okay, so exchange of views with uh, απόψε με την Επιτροπή σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την πρόοδο να αφορά τον πράσινο προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Jan Kodescu. Or not. Okay, Mr. Chair, instead of Mr. Jan Kodescu. <laughs> Mr. Jan Kodescu is replaced himself too? I'm, re I'm replacing Mr. Jan Kodescu. Τον εκπρόσωπο εγώ, ναι, απουσιάζει. Μα ο ίδιος ε, ε, κάποιον άλλον αντικαθιστούσε και τώρα εσείς είστε η αντικαταστάτρια του αντικαταστάτου. Ωραία ιστορία αυτή. Σάρα Ζιέν. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις ε, σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δύο χρόνια περίπου μετά ε, την ε, δημοσίευση του 2017 για την περιβαλλοντική νομοθεσία έχουμε 28 αναφορές εκθέσεις για τις χώρες. Όπως γνωρίζετε, στόχο έχει να βελτιωθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία και η πολιτική αυτή να εντοπίσουμε τις αδυναμίες για να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αναδιαιτία γίνεται ανάλυση, διάλογος και αξιολόγηση. Στόχος δεν είναι να ε, αντικατασταθεί η διαδικασία προσφυγής, αλλά να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη ε, επιτόπου και είναι ένα εργαλείο διαλόγου ε, εκτός από τη χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή ε, περιβαλλοντική νομοθεσία για πολλούς και ποικίλου που διαφέρουν και πολλοί από χώρα σε χώρα αλλά και από τομέα σε τομέα της οικονομίας. Τα τελευταία δύο χρόνια Πολλές ε, χώρες έχουν κάνει διαβούλευση και διάλογο, ιδιαίτερα με βάση τα προβλήματα και τις ε, προκλήσεις που έχουμε εντοπίσει στις συστάσεις αναχώρα και στις εκθέσεις αναχώρα. Ε, η προστασία της φύσης, η προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα είναι δύο από αυτά. Εκτός από αυτή τη βασική ενημέρωση και τεκμηρίωση, έχουμε επίσης λανσάρει ένα νέο μέσον ε, μεταξύ ομοτήμων peer-to-peer που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κάνουν ανταλλαγή πραγματογνωμοσύνης για ένα συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους για να βελτιώνονται πάρα πολύ ε, και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα πάντα στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Αυτό το μέσο έχει αποδειχτεί αρκετά επιτυχημένο και έχουμε πάνω από 19 έργα αυτή τη στιγμή και πολλά ακόμα περιμένουν. Τώρα ολοκληρώνουμε τη δέσμη EIR για το 2019 και αναμένεται να εκδοθεί τέλη Μαρτίου. Και πάλι θα έχει τη μορφή της ανακοίνωσης ε, που θα συνοψίζει τα ευρήματα της εκθεσεις αναχώρα και ένα άλλο παράρτημα που θα είναι η βασική ενημέρωση και το, το, ιστορικό ας πούμε για να μπορεί ο καθένας να δει ε, πού βρισκόμαστε, πού ερχόμαστε και πώς εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία σε λεπτομέρειες. Η υποστήριξή σας, οι προτάσεις σας έχουν ήδη γίνει ε, στην πρώτη φάση και ήταν πολύ σημαντική για να προετοιμάσουμε τη δεύτερη φάση αυτή το 2019. Οι νέες εκθέσεις καταγράφουν την πρόοδο που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη ή τη μη πρόοδο καμιά φορά. Και επίσης καλύπτουμε και νέα θέματα και νέους τομείς σε σχέση με το 2017. Κλιματική αλλαγή, χημικά, ε, βιομηχανικά στοιχεία ή νέα ε, χωροκατακτητικά είδη. από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις αναφοράς, αλλά ε, δεν υπάρχουν πάντα ε, οι ίδιες διαδικασίες, οι ίδιες προθεσμίες. Γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να τα ενοποιήσουμε κάπως. Και η νέα ανακοίνωση ε, θα αναφέρεται περισσότερο στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση με βάση μια μελέτη που θα εκδοθεί και αυτή το Μάρτιο αυτό θα βοηθήσει τις χώρες να συνεργάζονται, να έρθουν πιο κοντά και να εφαρμόζουν καλύτερα όλη αυτή την νομοθεσία. Τώρα προχωρώ στο πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η ένταξη της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των άλλων πολιτικών είναι υποχρέωση που απορρέει από τις συνθήκες για να έχουμε μια βιώσιμη κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να αποδίδει αυτό για να έχουμε κάποια συνοχή στις ευρωπαϊκές επενδύσεις με ε, μεταρρυθμίσεις. Η ετήσια ε, έκθεση για την ανάπτυξη του 2019 λέει ότι θα πρέπει στοχευμένες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, να συμβαδίζουν με πολύ καλά σχεδιασμένες ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις για να επιτύχουμε το στόχο μας προς μια κυκλική οικονομία ε, με μεγάλη μακροπρόθεσμη εφορία και μακριά από το διοξείδιο του άνθρακα. Ιδιαίτερα γίνεται λόγος για τις επενδύσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα για να προωθηθεί η παραγωγικότητα με μείωση του κόστους θα πρέπει να συνεχίσει η οικονομική ανάπτυξη να απαγκιστρώνεται, να αποσυνδέεται από τους ενεργειακούς στόχους για να φτάσουμε στους στόχους σύμφωνα με τις δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει και από τη Συμφωνία των Παρισίων. Άρα χρειάζονται επενδύσεις σε μια κυκλική οικονομία χωρίς διοξίδιο του άνθρακα με καινοτομία για να παραμένει η Ευρώπη ανταγωνιστική και να αυξηθεί η παραγωγικότητα χωρίς να κινδυνεύουν ε, οι συνθήκες διαβίωσής μας οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές θα πρέπει να ε, εξυγχρονιστούν για μια νέα μορφή κινητικότητας μετακινήσεων μέχρι και τις μηδενικές εκπομπές. Ε, χρειάζεται να διευρυνθεί περισσότερο το ενδεχόμενο και η δυνατότητα ιδιωτικών επενδύσεων με τοπικές ε, δράσεις και πρωτοβουλίες για να ξεφύγουμε από το διοξίδιο του άνθρακα και να μεταβούμε σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Τέλος, η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη λέει ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες μεταρρυθμίσεις και υπάρχει σαφής ε, συνέργεια ανάμεσα στη χρηστή διαχείριση, συγγνώμη, και την καλή λειτουργία των κρατικών μηχανισμών. Οι μελλοντικές προγραμματικές ε, αποφάσεις για το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να συνδέονται με όλα αυτά και με τις ανάγκες για επενδύσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζουρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν κατά τη διάρκεια όλης της παρέμβασης της Κομισιόν. Άκουσα όμως ένα τμήμα της. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δημιουργήθηκε ως εργαλείο οικονομικής συνεργασίας καταρχήν. Η τάση ήταν να διευρυνθεί σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, διαστάσεις και να μην ε, αποτελεί μόνο οικονομικό εργαλείο περιβαλλοντικές πολιτικές ε, είναι ε, συμπληρωματικές της οικονομικής συνεργασίας ε, για την, για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Εγώ έκανα διάφορες προτάσεις οι οποίες θα ψηφιστούν εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Πρότεινα την ε, δετερότητα του άνθρακα μέχρι το 2050 ως ε, στόχο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει στόχο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και επίσης πρότεινα στα, στα εθνικά προγράμματα ενέργειας που ε, τη χάνουν διαπραγμάτευση να περιλαμβάνονται και οι εθνικοί στόχοι ε, για την ενέργεια. Έτσι μόνο το ευρωπαϊκό εξάμεινο μπορεί να γίνει, να αποκτήσει και κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και να μην αποτελεί απλώς ε, μια οικονομική δέσμευση. Κανείς άλλος θέλει το λόγο. Ωραία, εγώ ίσως να κάνω μια ερώτηση. Πώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Mm. Σε σας ο λόγος. Thank you, Mrs. Είμαι επικεφαλής προϊστάμενος της, του τμήματος που συντονίζει ε, την εφαρμογή της μελέτης στο ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, θίξατε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε κανόνες χωρίς την εμπλοκή τοπικών και περιφερειακών αρχών. Προσπαθούμε να συμμετέχουν στο διάλογο με την βοήθεια της Επιτροπής των Περιφερειών διοργανώσαμε διάλογο και με τα κράτη-μέλη και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να φέρουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στο τραπέζι του διαλόγου. Επίσης, διεξάγουμε ανταλλαγές καλών πρακτικών και αλληλοεκπαίδευσης. Στηρίζουμε ε, με πόρους αυτή τη διαδικασία. Χρηματοδοτούμε, με άλλα λόγια, αυτή την ανταλλαγή εμπειριών, ε, τους εμπειρογνώμενες στη βάση δεδομένων κλπ. Και εκεί προφανώ περιλαμβάνεται και το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και μάλιστα διοργανώθηκαν στα κράτη-μέλη ε, και πολλά σημαντικά events, πολλές σημαντικέ εκδηλώσεις στι στις οποίες συμμετείχαν φορείς της ε, από τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. Βέβαια, όλα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη. Το πώς δηλαδή θα βοηθήσουν έτσι ώστε ε, να δοθεί και μια τοπική περιφερειακή διάσταση. Uh? Κύριε Σορίνιο, θέλετε ξανά το λόγο, όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες της Κομισιόν. Εδώ κλείνουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.